Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να καλωσορίσω στη συνεδρίασή μας την κυρία Ντανιέλ Νούι, την πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, στα πλαίσια του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού θεσπίστη, ε, ε και θεσπίστηκε το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Και μάλιστα όπως προβλέπει ο κανονισμός ε, και η διοργανική συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα έχουμε τακτικές ανταλλαγές απόψεων. Η πρώτη έγινε τον Ιούνιο και ελπίζω να έχουμε ανοιχτές, αποτελεσματικές και διαφανείς διοργανικές σχέσεις. Σήμερα περιμένουμε από εσά μια ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις ε, στον τραπεζικό τομέα και στην τραπεζική εποπτεία μετά ε, τις προσωμιώσεις ακραίων καταστάσεων, τι γίνεται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα MPLs, αλλά και ποια είναι τα μέτρα που εξετάζει η Επιτροπή Βασιλείας στα πλαίσια της ε, ε, εξεκέλευτης μεταρρύθμισης στον τραπεζικό τομέα. Θα ψηφίσουμε αύριο αυτό το θέμα. Γι' αυτό και περιμένουμε με ανυπομονησία την ενημέρωση που θα μας κάνετε. Μετά την εισαγωγική σας ομιλία θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που επανέρχομαι στην Επιτροπή σας για, σας, για να σας ενημερώσω και να ανταλλάξουμε απόψεις για την τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ. Πολλές αξιοσημείωτες εξελίξεις έλαβαν χώρα στον τραπεζικό τομέα και στην ενιαία ευρωπαϊκή εποπτεία από την τελευταία μου ακρόαση εδώ στην ΕΚΟΝ τον Ιούνιο και θα αναφερθώ σε αυτές πριν περάσουμε στις τελευταίες ε, μεταρρυθμίσεις της Επιτροπής της Βασιλείας και του Πλαισίου της Βασιλείας ε, όπως μου ζητήσατε. Ε, μεταξύ των βασικών ε, εξελίξεων στο τραπεζικό τομέα, η κερδοφορία των ε, τραπεζών της Ευρωζώνης είναι χαμηλή με βάση τα ιστορικά κριτήρια και η μέση απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης είναι 5,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2016, λίγο χαμηλότερο από το τέλος του 2015 που ήταν 6,5% αλλά διπλάσιο από αυτό του Δεκεμβρίου του 2014. Πάντως το να ε, ε, αποδίδουμε την ευθύνη για τη χαμηλή κερδοφορία στα χαμηλά επιτόκια δεν ε, είναι σωστό. Γιατί ήταν ανάμεικτα τα αποτελέσματα των χαμηλών επιτοκίων. Βέβαια, αρνητικά επηρεάζουν τα περιθώρια επιτοκίων, αλλά μετριάζουν τις πιστοτικές ζημίες και, στηρίζουν την αύξηση της πίστοσης και γενικώ ε, στηρίζουν και την ανάκαμψη της Ευρωζώνης, ε, βελτιώνοντας ε, το τραπεζικό κλίμα. Ε, σε αυτή τη συγκυρία έχουμε πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία. Για παράδειγμα, ο ανταγωνισμός από μη τραπεζικά ιδρύματα, αυξανόμενη ανάγκη σε επενδύσεις στην, στη τεχνολογία της πληροφορίας, ώστε να ανταποκριθούν οι τράπεζες στη, στη ζήτηση των καταναλωτών για ψηφιακές υπηρεσίες και ε, εξυγχρονισμό των διάβλων διανομής. Επίσης θα πρέπει να προσαρμόσουν και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Βέβαια δεν απόκειται στις εποπτικές αρχές να υπαγορεύσουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα ή να θέσουν στόχους κερδοφορίας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ίδιες οι τράπεζες θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο μακροοικονομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη πρόκληση στην ε, Τράπεζε αποτελούν τα MPL, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν αυξηθεί αισθητά από το 2008 και ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που χρειάστηκε να ακολουθήσουν προγράμματα ε, οικονομικής προσαρμογής και που ακόμη πασχίζουν να επανέλθουν στην ανάκαμψη. Συνεχίζουμε λοιπόν στην εκτό έργο, προσπαθώντας να υιοθετήσουμε μια συνεπή προσέγγιση για την εξηγίαση των μη εξυπηρετουμένων δανείων σε ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση. Όπως σας έχω πει και γραπτός, ε, ο ενιαίος ε, Εποπτικός Μηχανισμός έχει ε, ιδρύσει μια ειδική task force για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μετά από δημόσιες διαβουλεύσεις ε, θα καταλήξει σε κατευθυντήριες γραμμές για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα τελειώσουν το 15 Νοεμβρίου και εκεί θα αποκρισταλωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές κατά τον Ιανουάριο του 2017. Βέβαια, η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων ε, υπερβαίνει την εντολή των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ. Ε, γι' αυτό ε, απευθύνουμε έκκληση στο, σε όλους του ενδιαφέροντε ε, να άρουν τα διαρθρωτικά εμπόδια που εμποδίζουν τις τράπεζες να εξηγιάνουν τα κόκκινα δάνεια και να, να ε, διευκολύνουν μια αναδιάρθρωση αυτών των καθυστερούμενων δανείων. Επίση, χρειάζεται ένα εξορθολογισμό των πλαισίων αφαιρεγκαιότητα και των σχετικών διαδικασιών στα κράτη-μέλη. Τώρα, για την διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγηση, ΣΡΕΠ 2016. Το εγχείρημα αυτό αποκάλυψε ότι το επίπεδο κινδύνου στο σύστημα είναι σχετικά σταθερό, αλλά οι τράπεζε τη Ευρωζώνη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάφορε προκλήσει. Ήδη ανέφερα την κερδοφο κερδοφορία, τη χαμηλή κερδοφορία και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και μάλιστα σε μερικέ τράπεζε θα πρέπει να τεθούν και ζητήματα διακυβέρνηση. Επίση, τα εποπτικά τεστ, ε, stress test έδειξαν κάποιε ευπάθειε ε, στου δυσμένου κραδασμού. Όπω είπα και στην ακρόαση του Ιουνίου, και μετά από πολλέ διευκρινήσεις που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ερμηνεία τη κοινοτική νομοθεσία, θα εκφράσουμε τις εποπτικές μας προσδοκίες για τα κεφάλαια φέτος ε, στα πλαίσια των απαιτήσεων του δεύτερου πυλώνα και των κατευθυντηρίων γραμμάτων του δεύτερου πυλώνα. Και μάλιστα το συνολικό, συνολικό κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1 θα, θα παραμείνει σχετικά σταθερό σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που διαπιστώσαμε κατά τη δεύτερη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγηση, που έγινε στα πλαίσια των εποπτικών αρμοδιοτήτων τη ΕΚΤ ήταν πόσο σημαντική είναι η εποπτική κρίση κατά τη θέσπιση του δεύτερου πυλώνα με εναρμονισμένο και συνεπή τρόπο για όλα τα σημαντικά ιδρύματα και οργανισμού. Ε, δεν θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τους ειδικού κινδύνους ε, με μονομένων επιχειρηματικών μοντέλο... χρησιμοποιώντα μόνο μία αμυγός ε, μηχανιστική προσέγγιση τύπου πυλώνα 1 με μία ενιαία αντιμετώπιση. Ε, γιατί μία ειδικευμένη, εξατομικευμένη προσέγγιση αναγνωρίστηκε και από το κανονισμό μετά την κρίση ε, που πρότεινε στους ε, Ευρωπαίους επόπτες ε, την επιβολή απαιτήσεων ανάλογα με τον κίνδυνο στα πλαίσια του πυλώνα 2. Και αυτό θα διαφυλαχθεί στην επερχόμενη αξιολόγηση και αναθεώρηση ε, του τραπεζικού κανονισμού. Τώρα, να δούμε τι μεταρρυθμίσεις εξετάζει η Επιτροπή της Βασιλείας. Καταρχήν, ε, η υπερβολική αστάθεια στον υπολογισμό ε, των κινδύνων των εσωτερικών προτύπων υπονομεύει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου, του κεφαλαϊκού πλαισίου της Βασιλείας και δημιουργεί ανασφάλεια για τους τραπεζικούς επενδυτές. Και οι επόπτες και οι αγορές συμφωνούν ότι ε, δεν μπορούμε όλες τους τραπεζικούς πιστοτικούς κινδύνους να τους, ε, ε, σε τους υπαγάγουμε σε συγκεκριμένα πρότυπα. Αναγνωρίζοντας αυτά τα προβλήματα, λοιπόν, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέτασε και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Για παράδειγμα, ε, αναθεώρηση των ε, εσωτερικών αξιολογήσεων των πιστοτικών κινδύνων, περιορίζοντας ε, τα πρότυπα για συγκεκριμένους κινδύνους ή καταργώντας αυτά τα πρότυπα για εκθέσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για ακριβείς εκτιμήσεις. Και μάλιστα η Επιτροπή τη Βασιλεία εξετάζει και διαφορετικέ προσεγγίσεις για την οριστικοποίηση αυτών των αναθεωρήσεων. Μία αναθεώρηση τη της τυποποιημένη προσέγγιση για το πιστοτικό κίνδυνο, με βασικό κίνδυνο να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ τη ευαισθησία στον κίνδυνο και τη απλότητα, και μία αναθεώρηση του πλαισίου για τον επιχειρηματικό κίνδυνο, με συμπερίληψη τη ε, πιθανότητα αντικατάσταση του παρόντο προτύπου με μία νέα προσέγγιση τυποποιημένη και ευαίσθητη στον κίνδυνο όπου θα χρειαστεί, θα γίνουν κάποιες προσαρμογές στα πλαίσια μετά από διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις αυτές συνεχίζονται για την καταλληλότητα ενός κατώτατου ορίου κεφαλαίου στα εσωτερικά πρότυπα με βάση τις αναθεωρημένες τυποποιημένες ε, προσεγγίσεις. Ταυτόχρονα οι τελικές ε, τροποποίησεις στο συντελεστή μόχλευσης ε, ήδη γίνονται και είναι σημαντικές για να γίνει η στάθμιση του του πιθανού, της πιθανής επιβάρησης των συστημικών τραπεζών και να εξασφαλίσουν ε, ότι η έκθεση στα μέτρα καλύπτει ε, κατάλληλα τις σχετικές δραστηριότητες. Η αναζήτηση της σωστής ισορροπίας μεταξύ της ευαισθησίας των κίνδυνο και της απλότητας δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να αντιληφθούμε και ότι και η αλλαγή της πολιτικής συμβάλλει σε κάτι τέτοιο και η μείωση της δικαιολόγητης αστάθειας, αλλά και ο αντίκτυπο που έχουν οι αλλαγέ ε, στι δικαιοδοσίε. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη για να έχουμε ένα ισορροπημένο πακέτο. Τώρα, να δούμε το ρόλο της ΕΚΤ. Ε, η ΕΚΤ θεωρεί πολύ σημαντικό αυτό το έργο και ε, έχει συναντήσεις ε, πριν τις συνεδριάσεις με εκπροσώπους της Ευρωζώνης για να εξετάσει αυτά τα θέματα στις χώρες του ενιαίου οπτικού μηχανισμού. Και γενικώ σε επίπεδο βασιλεία η ΕΚΤ συμμετέχει ενεργά στο τεχνικό έργο για τις ε, μελέτες επιπτώσεων. Ελπίζουμε ε, Τη Επιτροπή Βασιλεία για την Τραπεζική Εποπτεία. Είναι σημαντικό να η τελική στάθμιση αυτών των μεταρρυθμίσεων να μην καταλήξει υπερβολική αύξηση των κεφαλαϊκών απαιτήσεων, όπως είχαν υποσχεθεί τον, ε, Ιούνιο, τον Ιανουάριο του 2016 και επανέλαβαν τον Σεπτέμβριο του 2016 οι διοικητέ κεντρικών τραπεζών και επικεφαλής ε, εποπτικών αρχών. Αυτό επιβεβαιώνεται και πάλι. Τώρα, είναι πολύ πρόωρο να προεξοφλήσουμε την έκβαση σε αυτό το στάδιο. Σε ό,τι αφορά την τιτλοποίηση, χαιρετίζουμε τι αρχικέ προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί βρίσκω τη σωστή ισορροπία μεταξύ τη ανάγκη να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή αγορά τιτλοποίηση και τη ανάγκη ε, να διατηρηθεί ο προνοητικό χαρακτήρα ε, του κανονιστικού πλαισίου. Η τιτλοποίηση μπορεί να συμβάλλει σε μια καλά διαφοροποιημένη χρηματοδοτική βάση για τι τράπεζε και μάλιστα στην παρούσα συγκυρία, όπου υπάρχουν περιορισμοί στα κεφάλαια των τραπεζών, ε, θα είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε μια εύρυθμη αγορά τιτλοποίησης. Επίση, καλά σταθμισμένοι ε, κανονισμοί χρειάζονται. Και οι δύο νομοθετικές ε, πράξεις αποφεύγουν τα λάθη του παρελθόντο που οδήγησαν στη χρηματοπιστωτική κρίση και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν ότι οι ευρωπαϊκές αγορές τιτλοποίησης που ήταν σχετικά ασφαλείς κατά τη διάρκεια τη κρίση, θα αναζωογονηθούν με υπεύθυνο τρόπο. Θα ήθελα εν κατακλείδη να διαπιστώσω ότι σημειώνουμε αρκετή πρόοδο σε πολλά θέματα που είναι ζωτική σημασία για την Τραπεζική Ένωση, όπως ε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά θα χρειαστούν ε, περαιτέρω προσπάθειες που θα πρέπει να συμπληρωθούν από ρυθμιστικέ δράσεις αλλά και πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η ε, τραπεζική εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κέντρική Τράπεζας είναι έτοιμη και πρόθυμη να σας παράσχει υποστήριξη. Και Ευχαριστώ για την προσοχή και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ και φυσικά και η Επιτροπή μας θα συμμετάσχει και θα σχολιάσει όλα τα ζητήματα που αναφέρεται. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Brian Hayes. Κύριε Νουή, ε, καλώς ορίσατε ξανά στην ΕΚΟΝ και ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Είχαμε μία συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών τον περασμένο μήνα όπου τέθηκε το ζήτημα των NPL των μη εξυπηρετούμενων δανείων που επισημάνατε και εσείς σήμερα και επί τη ευκαιρία εκείνη ο κύριος Ενρία είπε ότι τα 13 κράτη-μέλη κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια άνω του 5%, σε ποσοστό άνω του 5%, τα περισσότερα από αυτά ε, κράτη τη Ευρωζώνη. Και έτσι ξεκίνησε μια διαβούλευση ε, και καθοδήγηση προ τι τράπεζε Το καλωσορίζουμε. Στη δική μου ε, χώρα, στην Ιρλανδία, το ποσοστό αυτό είναι 14% των NPL. Είναι υπερβολικά υψηλό. Παρότι έχει πέσει από το 19% και σημειώθηκαν καποιέ βελτιώσει ειδικότερα από εμπορική άποψη περισσότερο παρά από λιανική. Ε, είναι σημαντική αλλαγή αυτό για τις τράπεζες. Να σας ρωτήσω, από ρυθμιστική άποψη, τι συμβολή θα δίνατε στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής στην Ιρλανδία και στους διευθυντές τραπεζών για το πώς θα μπορούσαν να επιλύσουν τα έκρεμοντα ζητήματα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ειδικότερα εκείνα που έχουν διάρκεια μεγαλύτερων δύο ετών. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις Επίσης αναφερθήκατε σε διαρθρωτικά εμπόδια, δομικά εμπόδια. Ποια είναι η προτεραιότητα κατά την απόψή σας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και τέλος για το Βασιλεία που συζητείται εκτενώς σε αυτήν εδώ την Επιτροπή όπως τα γνωρίζετε. Η ανησυχία είναι ότι θα καταλήξουμε σε κάποιο σκληρό εργαλείο ρυθμιστικό για την αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων ε, τι πιστεύετε θα ήταν το σωστό αποτέλεσμα. Πώς θα επιτύχουμε την ισορροπία που θέλουμε ώστε να αποκαταστήσουμε την ε, ε, εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, να έχουμε διαφάνεια και να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους και να τους εκτιμάμε και σωστά. Και, επι... ε, και τέλος, πώς θα επηρεάσει το αποτέλεσμα αυτό τα stress test που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σημερινού τραπεζικού καθεστώτος. Ευχαριστώ. Yeah. Uh, well, uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, όσον αφορά την κατάσταση των Ιρλανδικών τραπεζών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τη σχετική έκθεση. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμμετοχή των συναδέλφων σα για την αντιμετώπιση του ζητήματο. και όπω έχουν τα πράγματα, ο άνθρωπο που καθοδηγεί τις εργασίες μα είναι η Σαναντονορία από την Ιρλανδία, ε, αναπληρωτής ε, διευθύντρια της Κεντρικής Τράπεζας, γιατί η Ιρλανδία ακριβώ βρήκε κάποιε καλές λύσει και έχει σημειώσει καλή πρόοδο Οπότε κινούμαστε και προς την ίδια κατεύθυνση με τις ε, χώρες της Ευρωζώνης. Ε, συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την οποία αναφέρατε, η οποία εκπροσωπείται στην ομάδα εργασία της Αυτό είναι πολύ καλό. Πρόσφατα εκδώσαμε δύο έγγραφα και αναφερθήκατε στις κατευθυντήρες γραμμές που θα μπορούσαν να δοθούν στους υπευθύνους χαράξης πολιτικής, στους νομοθέτες. Έχουμε μία άσκηση απολογισμού όπου οκτώ χώρες ε, εξετάζονται για να δούμε την κατάστασή τους όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, πιθανά εμποδία για τη δημιουργία ε, επιχειρήσεων διαχείρισης ε, ε, περιουσιακών στοιχείων, γενικώ για τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε νομοθετήματα. Επτά χώρες έχουν υψηλό επίπεδο έκθεσης, μία χώρα όχι, αλλά εμείς θα εκδώσουμε έναν απολογισμό και για τις 19 χώρες και αυτό παρατηρούμε είναι ότι πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε σωστούς κανόνες χρεοκοπίας. Και εγώ ε, ελπίζω να ε, έχει καλό αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό έργο για την περίπτωση χρεοκοπιών ε, για τις επιχειρήσεις. Κάτι που θα είναι υποφελές και πέραν της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών. Ε, και για τους επενδυτές ε, που ενδεχομένως θα ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ε, μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα πρέπει να μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η νομική αντιμετώπιση και να δουν κατά πόσο ενδιαφέρονται ή όχι. Χρειαζόμαστε λοιπόν νόμους σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Και χρειαζόμαστε και δικαστήρια, δικαστές που να ε, εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες. Υπάρχουν πολλά είδη μη εξυπηρετούμενων δανείων ε, εταιρικά, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ατόμων για τα πρόσωπα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες ε, διαδικασίες κατεπήγοντος με ειδικού δικαστές και επίσης και εξοδικαστικές λύσεις θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή. Οι περισσότερε χώρε που έχουν αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα κινούνται προ αυτή τη σωστή κατεύθυνση. Στη Γαλλία ξεκινήσαμε όπως και στην Ιρλανδία με την ποιοτική καθοδήγηση για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Έχουμε και άλλη μια φάση παράλληλη που είναι η κοινή υποπτική ομάδα που διεξάγει εποπτικό διάλογο με τις τράπεζες, ε, εποπτεί, δηλαδή εποπτεύει ώστε να βεβαιώνεται ότι κινούνται οι τράπεζες προς σωστή κατεύθυνση με ταχύτητα που μπορούν φυσικά, γιατί δεν μπορούν όλες οι τράπεζες να κινηθούν με την ίδια ταχύτητα. Είμαστε φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστές. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την κατάσταση της εκάστοτε τράπεζας, του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου της εκάστοτε χώρας. Τώρα, όσον αφορά τον κίνδυνο των ε, ε, σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων που θα προκύψει από την ε, μεταρρυθμίση της Βασιλείας. Ποιο θα ήταν ε, το, ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, το να υπάρχει συμμόρφωση με την εντολή που παρήχε ο οργανισμός αναφοράς της Επιτροπής Βασιλείας, δηλαδή μη σημαντική με ένα αυξή κεφαλαίου αλλά διορθώσεις Αυτές είναι οι πρώτες προσδοκίες. Και θα πρόσθετα το εξής, το να υπάρξει μια τυποποιημένη προσέγγιση ικανοποιητική που θα εξετάζει τους, την πολυμορφία των κινδύνων. Αν υπάρχει λοιπόν μια τέτοια τυποποιημένη προσέγγιση θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι καλής ποιότητας. Μπορεί μάλιστα να σε ορισμένες τράπεζες που ενδεχομένως δεν ε, έχουν περιθώριο να δαπανίσουν πολλά χρήματα στην οικοδόμηση μοντέλων και στη διατήρησή τους. Μπορεί να τους οθήσει λοιπόν να καταφύγουν σε αυτές ε, τις απλές ε, αλλά προσαρμοστικές τυποποιημένες προσεγγίσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Πρεβανς Ευχαριστώ για τη Βασιλεία 3. Γιατί αυτό το θέμα μας αποσχολεί ιδιαίτερως, να έχουμε και μια ευρωπαϊκή φωνή, κυρίως την φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πρέπει να εισακουστεί πριν ολοκληρώσει η Επιτροπή Βασιλείας το έργο της σε αυτή τη φάση. Θα ήθελα λοιπόν να εξακριβώσω ποια είναι τα βασικά μηνύματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τη δική σας γνώση του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος και τον εντοπισμό των κινδύνων που κάνατε Ποια κατά τη γνώμη, είναι τα είναι τα βασικά μηνύματα που θα πρέπει να δώσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ε, ε, Επιτροπή της Βασιλείας για να ληφθούν υπόψη και η δική σας, ε, και η δική σας ανησυχία. Και ένα ζήτημα βασικής σημασίας που βρίσκεται στο επίκεντρο των εργασιών της Βασιλείας ε, και εκεί έγκυται η διαφορά μας με τους Αμερικανούς που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη προσέγγιση ενώ οι δικές μας τράπεζες με μεγέθου χρησιμοποιούν τα εσωτερικά πρότυπα αξιολόγηση. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Και φυσικά θα πρέπει πρώτα για να εισακουστεί η φωνή μας να είναι ενιαία και ηχηρή, κάτι που δεν είναι αυτονόητο ή αυτόματο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαπραγματεύσει αυτές είναι πολύ σοβαρέ και δύσκολε όπω διαπιστώσαμε. Και γι' αυτό αναδύεται η ανάγκη ε, να αποφαινόμαστε με μία ενιαία φωνή και να μην υπάρχει διάσπαση των προσπαθειών. Και το πλονέκτημα του ενιαίου αποπτικού μηχανισμού είναι ότι δίνει φωνή σε πολλές χώρες που δεν κάθονται στις διαπραγματεύσεις στην Επιτροπή Βασιλείας, αλλά είναι μέλη του εποπτικού, ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Εν τη λοιπόν. Επίσης είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε συμφωνία δεν ενθαρρύνουμε τις τράπεζες ε, να δηλώνουν ότι καλύτερα καμία συμφωνία ε, από ότι μια κακή συμφωνία. Θέλουμε μια καλή συμφωνία για όλους μας ε, και για μας και για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Και φυσικά γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τραπεζικών συστημάτων δεν είναι θέμα αντιπαράθεση με τι Ηνωμένε Πολιτείε ή αντιπαράθεση των μοντέλων του τυποποιημένου από τα πρότυπα εσωτερική αξιολόγηση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση των προσωμιώσεων ακραίων καταστάσεων, που ε, και αυτά τα stress test πρότυπα είναι. Δεν γίνονται ποτέ προσωμιώσει ε, ακραίων καταστάσεων χωρί μοντέλα, χωρί πρότυπα. Ενώ εμείς χρησιμοποιούμε τα πρότυπα που έχουμε στα ευρωπαϊκά κείμενα ή στα κείμενα της Επιτροπής της Βασιλείας. Αυτό που χρειάζεται είναι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, ο SSM, να κάνει μια της ποιότητας των μοντέλων και μάλιστα συνεκτική και συνεπή στις 19 χώρες. Γιατί πριν τον ενιαίο αποπτικό μηχανισμό, πολλά πράγματα γίνονται με διαφορετικό τρόπο στι 19 χώρε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σωστή ε, κύρωση και διακρύβωση των μοντέλων και στη συνέχεια να αναγκάζουμε τις τράπεζες να τα εφαρμόζουν με σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο. Τότε θα είμαστε και αξιόπιστοι στο διάλογο. Πολλά πράγματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γίνεται, για παράδειγμα, λόγος ε, για την αντιμετώπιση των ανυπόθηκων δανείων στις συζητήσεις στην Επιτροπή Βασιλείας. Ε, ενώ στις Αμερικανικές τράπεζες, στους λογισμούς των Αμερικανικών τραπεζών δεν έχουμε πολλά τέτοια ενυπόθηκα πια δάνεια. Το μήνυμά μας πάντως θα πρέπει να είναι αξιόπιστο απέναντι στους Αμερικανούς. Δεν είμαι απεσιόδοξη ως προς την έκβαση των διαπραγματεύσεων, γιατί και καλή εκπροσώπηση έχουμε και το ρόλο μας διαδραματίζουμε πλήρως. Ο κύριος Λόπες Βερμέχο. Η κυρία Λόπες Βερμέχο, συγγνώμη. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας και ευχαριστούμε την κυρία Νουή για την παρουσία της. Στις τελευταίες προσωμιώσεις ακραίων καταστάσεων δεν έλυθησαν υπόψη πολλοί κίνδυνοι που ε, επηρεάζουν την τράπεζα και χρησιμοποιήθηκαν κάποιες ε, ε, βαθμονομή, κάποιε σταθμίσει ε, διαφανείς. Δεν εν υπόψη το Brexit, η δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τον κίνδυνο να δημιουργηθούν νέε φούσκε εξαιτία του προγράμματο τη ποσότική χαλάρωση. Δεν λήφθησαν υπόψη νέοι κίνδυνοι συγκέντρωση και τραπεζική συγκέντρωση και τραπεζική ρυθμίση. και μάλιστα το γεγονό ότι ε, παρα, παραλύθηκαν κάποιες σημαντικές τράπεζες ε, με προβλήματα φεραγιότητα κάποιων χώρων, διακυβεύει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Ε, είναι οικουμενικό το πρόβλημα με, τις, ε, με τα stress test που δεν λαμβάνουν υπόψη επαρκώς όλους τους κινδύνους. Γιατί λοιπόν παραλαμβάνετε αυτό το λάθος. Επίσης ως προς την ανεξαρτησία του έργου σας. Σήμερα έλαβα την απάντησή σας ε, σε μια γραπτή ερώτηση που είχα κάνει για την Deutsche Bank και το μικροσκάνδαλο που έγινε με την αγορά του URG γιατί ε, έχετε αυτή την πληροφορία και όχι αγοραπολίσεις άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων. Μήπως έγινε μια χειραγώγηση των αποτελεσμάτων τόσο σημαντικής τράπεζας, τόσο συστημικής τράπεζας όπως είναι η Deutsche Bank. Στην πρώτη σας γραπτή απάντηση μου είπατε ότι οι προσωμιώσεις ακραίων καταστάσεων δεν έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογούν τους συστημικούς κινδύνους. Ρωτώ λοιπόν, αν τα stress test δεν μπορούν να αξιολογήσουν το συστημικό κίνδυνο μιας νέας ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης κατάρρευσης, προς τι τότε τα stress test. Σε ό,τι αφορά τη Βασιλεία, συμφωνείτε να μειωθούν οι κεφαλαϊκές απαιτήσει για τις συστημικές αυτές τράπεζες. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Λέτε ότι τα stress test ε, δεν λαμβάνουν υπόψη τα, στα σενάρια τους όλους τους κινδύνους που μπορεί να διατρέξει μια τράπεζα. Ναι, έχετε δίκιο. Τα stress test ε, δεν προβλέπουν ε, την οικονομική χρηματοπιστωτική κατάσταση. Πρέπει να είναι στοχευμένα σε συγκεκριμένους κινδύνους ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να εξάγουμε τα ε, κατάλληλα συμπεράσματα. Δεδομένων αυτών, να σας υπενθυμίσω ότι ο ενέος μηχανισμός υποπτίας δεν αποφάσισε για τα σενάρια των stress test, τα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Εμείς δεν έχουμε λόγο και επίσης η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών χρησιμοποιεί ε, πολλές ε, απόψεις πολλών ε, συμμετεχόντων για να αποφασίσει τα σενάρια. Για παράδειγμα, προβλέψεις της Κομισιόν για τα βασικά σενάρια, η εκτίμηση κινδύνου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικών Κινδύνων, η SRB, το οποίο επίσης ε, συνεργάζεται με την Γενική Διεύθυνση Financial Stability της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δεν είναι Γενική Διεύθυνση του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας οπότε πιθανότατα εμείς στην SSM είμαστε πιθανότατα οι μόνοι που δεν ε, καθορίζουμε τα σενάρια και πιστεύω ότι σωστά είναι τα πράγματα έτσι γιατί αλλιώς θα υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων οπότε παίρνουμε τα σενάρια ως δεδομένα και βάσει αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε καλύτερα. Πιστεύω ότι το ESRB ε, ε, ειδικότερα παρέχει αυτή τη μακροοικονομική ρεαλιστική διάσταση που αναφέρατε. Η δυσκολία φυσικά ε, έγκυται στο γεγονός ότι στις 28 ευρωπαϊκές χώρες σε καθεμία από αυτές η κατάσταση είναι διαφορετική όσον αφορά την, ε, μακρο, το μακροπροληπτικό τοπίο και την κατάσταση. Ε, ταυτόχρονα όλες οι χώρες και όλες οι τράπεζες χρειάζονται μακροπροληπτική πολιτική ε, και τα σχετικά εργαλεία. Αλλά ακριβώς τα stress τα σενάρια στα οποία βασίζονται ε, αφορούν τη μακροοικονομική κατάσταση. Τώρα όσον αφορά τα stress test ε, συμφωνώ ότι ορισμένε φορές πρέπει να ε, επανασχεδιάζουμε τα stress test. Χρησιμοποιούμε τις ίδιες μεθόδους εδώ και αρκετό καιρό και Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, να συνεργαστούμε για να κενήσουμε τη μεθοδολογία του εγχειρήματο αυτού. Ε, η επόμενη έσκηση θα είναι όχι του χρόνου, ε, σε δύο χρόνια. Αυτή είναι η περιοδικότητα. Μου λέτε... Αναφερθήκατε στην Deutsche Bank. Εγώ διαφωνώ μαζί σας. Ξέρετε, η βάσει της μεθοδολογίας του stress test ε, ε, ε, αναφερόμαστε σε στατικό ισολογισμό, δηλαδή κάθε χρόνο οι τραπεζές υποτίθεται κάνουν το ίδιο πράγμα, τα ίδια λάθη κατά επανάληψη, τα οποία δεν θα, γεγονός δεν θα συνέβαινε στην πραγματικότητα, Οπότε, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν παρεκκλήσεις κατά την άσκηση stress test. Αν πάρουμε δυναμική εξισορρόπηση, ε, ε, συγγνώμη, ε, δυναμικ, δυναμικούς ισολογισμούς, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά όταν έχουμε στατικό ισολογισμό, εκεί αναθεωρούμε ε, τα πράγματα βάσει συγκεκριμένων ετοιμάτων από τις τράπεζες. Το καλύτερο, ξέρετε, είναι να πούμε το πιο άνετο, το πιο εύκολο, να πούμε όχι στα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι πιο εύκολο. Ξέρετε, μερικές φορές και εγώ ε, τίνω να θέλω να πω κάτι τέτοιο, αλλά όταν έχουμε μια δύσκολη κατάσταση εποπτείας, ε, εξετάζουμε τις περιπτώσεις ε, που μας υποβάλλονται ουσιαστικά και τέτοια ήταν η περίπτωση της Deutsche Bank. Μάλιστα υπήρχε και άλλη μία που δεν είχε συμπεριληφθεί στην, ε, στο stress test της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αλλά στη ΣΡΕΒΑ όπου δύο τράπεζες αντιμετωπίστηκαν με τον ίδιο τρόπο. Το εγχείρημα λοιπόν ε, ολοκληρώθηκε. Ε, ε, συμπεριλήφθηκε στους λογαριασμούς του 2015 της Deutsche Bank που ελέγχθηκε από ορκωτούς λογιστές και πράγματι η άδεια της Κινέζικης Εποπτικής Αρχής δεν είχε καν δοθεί, αλλά ανάλογα με τις εθνικές νομοθεσίες μπορεί να δοθεί πριν ή μετά σε, μεγάλες τέτοιες, ε, σε μεγάλα τέτοια εγχειρήματα προηγούνται κάποιες επαφές ε, ώστε να μην σπαταλάτε χρόνο σε περίπτωση ένστασης. Είδαμε λοιπόν ότι είχαμε κάθε λόγο και εξακολουθώ να το πιστεύω ότι είχαμε κάθε λόγο να κάνουμε αυτό που κάνουμε πρόσφατα. Πρώτα απ' όλα όλα ήταν δημόσια. από την πρώτη μέρα. Όλο το υλικό που παρήχε, τίποτα δεν ήταν απόρριτο, όλοι μπορούσαν να πάνε να το δουν. Και ψηφίστηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο του SSM και το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΜΠΑ. Οπότε έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν πιστεύω ότι κάναμε κάτι λάθος. Και σίγουρα δεν αντιμετωπίσαμε την τράπεζα, την Deutsche Bank, διαφορετικά από τις άλλες τράπεζες. Ε, είναι λάθος μια τέτοια άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή την ετήσια ακρόαση και θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι η ατμόσφαιρα γενικά όταν μιλάμε για τον δημοσιονομικό κανονισμό αλλάζει πηγαίνουμε κατά των ισχυρότερων κανόνων αλλάζει ο τόνος και γενικά θέλω να πω πως είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχουμε το μηχανισμό ε, σταθερότητας. Ε, χωρίς αυτόν θα έλεγα πως έχουμε έναν ρυθμιστικό ανταγωνισμό προς τα κάτω. Και από ό,τι ακούω ε, κάνετε καλή δουλειά. Αυτό θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι δεν έχετε... Δεν είστε πλήρως ελεύθεροι από αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτά τα οποία έχουν συμβεί όσον αφορά την ε, μεταχείριση του NDA και τον διαχωρισμό των απαιτήσεων του πυλώνα 2 όσον αφορά τη την υποχρεωτική πτυχή του πυλώνα 2 δεν έχει βάση στο ευρωπαϊκό δίκαιο και νομίζω πως ανταποκριθήκατε σε πιέσεις και προχωρήσατε πέρα από τα συμφωνημένα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Τώρα, για τα stress test πρέπει να είμαστε σαφείς για την ε, Deutsche Bank. Οι κανόνες λένε πως μπορεί να γίνει μια εξαίρεση εάν η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί. Η συναλλαγή αυτή για την οποία έγινε εξαίρεση δεν είχε ολοκληρωθεί το 2015, επιβεβαιώθηκε από τις κινέζικες αρχές ε, ε, πολύ προσφάτως. Και άρα δεν ακολουθήσατε τους κανόνες. Γι' αυτό ακριβώς η EBA έκανε την εξαίρεση αυτή με ένα ερωτηματικό στις δημοσιεύσεις της για την Deutsche Bank. Θα ήθελα να μας πει τα πράγματα ξεκάθαρα γιατί δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τα τεστ ε, κοπόσεων των τραπεζών να μην είναι τα ίδια για όλα τα κράτη-μέλη και τις τράπεζες. Και ο λόγος μόχλευσης της Deutsche Bank φαινόταν ότι ήταν πάνω από το 3% παρά το ότι στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι παρακάτω. Και εκεί πέρα το γράμμα σας, ε, η επιστολή σας προς τον Φάμπιο Ντεμάζη δεν είναι ε, πιστικό και μάλλον δεν ακολουθείτε τους ίδιους σας τους κανόνες. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα συμφωνώ πλήρως με το γεγονός πως ο τόνος ε, του κανονισμού δεν θα πρέπει να αλλάζει στο μέτρο του δυνατού. Γιατί η σταδιακή εφαρμογή των νέων κανονισμών δεν έχει τελειώσει η εισαγωγή τους. Πρέπει να εφαρμόσουμε τους κανονισμούς και να δούμε το ότι από πού προέρχονται αυτοί οι κανονισμοί. Αυτά τα πράγματα λοιπόν χρειαζόταν και πρέπει να εφαρμοστούν. Ε, Αυτή είναι η στάση του, ε, του μηχανισμού στήριξης. Ε, δεν θέλουμε ακριβώς περισσότερες απαιτήσει στον πυλώνα 1. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να συμμορφωθούμε πλήρως με τις απαιτήσει ε, του ΓΚΑΣ. Όσον αφορά τις κατευθύνσεις του πυλώνα 2 για το μέγιστο ποσό διανομής, ζητήσαμε διευκρινήσεις από την ε, Κομισιόν γιατί οι νομικοί μας μας έλεγαν ότι υπήρχαν ε, διαφορετικές πιθανές ερμηνείες για το τι έπρεπε να γίνει. όσον αφορά την ε, κατάταξη των διαφόρων αποθεματικών. Ζητήσαμε λοιπόν αυτή την διευκρίνηση, μας την έδωσαν, έπρεπε να την εφαρμόσουμε. Ο στόχος είναι ότι οι απαιτήσει του πυλώνα 2 είναι οι κατευθύνσει του 2016 χοντρικά ισοδυναμούν με τι απαιτήσει του πυλώνα 2 τα προηγούμενα χρόνια γιατί είπαμε ότι είμαστε σε μια σταθερή κατάσταση. Οι κατευθύνσει ε, από τι εποπτικές αρχές είναι κάτι πολύ σοβαρό και αναμένουμε οι αρχές να συμμορφωθούν με αυτό αλλά δεν είναι η μέγιστη. Ναι, αλλά η συμβουλή της Κομισιόν και της CBA ήταν σκληρότερη από αυτό το οποίο κάνατε εσείς και δεν έχετε νομική βάση γι' αυτό. Όχι, εγώ δεν νομίζω. Bloomberg είπε, το είπε αυτό, λέει ο κύριος Γκίγκολτ και ήταν σαφές. Ε, ειλικρινά δεν νομίζω, είναι η απάντηση της κυρίας Νοή. Αλλά ευχαρίστω να συζητήσω τις λεπτομέρειες μαζί σας. Αυτό το κάναμε Αναφέρατε τις μεγάλες ε, τράπεζες. Η επιστολή από τις μεγάλες τράπεζες ήρθε το 2015, όχι το 2016. Και το εφαρμόσαμε ακριβώς αυτή την, ε, κα, τις κατευθυντήρες μας της EBA. Ε, Και θεωρούσαμε ότι η λύση αυτή, η εφαρμογή των διευκρινήσεων αυτών ήταν κάτι το οποίο θα γινόταν, αλλά δεν αφορά βεβαίω το μέγιστο ποσό διανομής, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται αυτόματα. Ξεκινάει ένας διάλογος, ε, κεφαλαιακές απαιτήσεις, ε, αναμένουμε την απάντηση της τράπεζας πριν λάβουμε κάποια εποπτικά μέτρα. Αυτή είναι η εξήγηση. Για το ότι δεν έχει σχέση με το μέγιστο ποσό ε, διανομής. Τώρα για την Deutsche Bank ε, την περίπτωσή της. Θεωρώ ότι κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε. Ε, είπατε πως έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση το 2015, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται άπαξ είναι στους λογαριασμούς, στον ισολογισμό της τράπεζας. Ακριβώς όταν δεν είναι σαφής η κατάσταση ε, γύρεται τέτοιο θέμα. Δεν είναι μόνο θέμα Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για, και απόφαση της CBA να αποκαλύψει τις πληροφορίες, αφορούσε και το, το μηχανισμό, τον εποπτικό μηχανισμό. Θέλαμε να είναι γνωστό δημοσίω. Δεν ξέρω, ίσως ήμασταν πολύ δίκαιοι και όχι αρκετά σκληροί. Ίσως έπρεπε να πούμε και κάποιο όχι. Αλλά μια φορά, εντάξει, ίσω να υπήρχαν και γελία αποτελέσματα. Γι' αυτό ε, εξετάζουμε πάρα πολύ σοβαρά τα ερωτήματα τα οποία μας θέτουν και αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίζαμε οποιαδήποτε τράπεζα στην ίδια κατάσταση με τον ίδιο τρόπο. Για να είμαστε δίκαιοι, θεσμικά, Λέω ο πρόεδρος, πρέπει να πω πως κάθε άποψη βεβαίω είναι δεκτή, αλλά βεβαίω είχε ψηφίσει και το Κοινοβούλιο με στόχο να μην υπάρχει ακριβώς αυτό το θέμα με τα μερίσματα για να είμαστε σκληροί σε αυτό το ζήτημα. Ε, από ό,τι κατάλαβα η δεν έχει πρόβλημα με αυτή τη λύση. Λοιπόν, Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τις απαντήσεις που μόλις δώσατε για την Deutsche Bank και όσον αφορά την αξιολόγηση στα τελευταία stress test τα 4 δισεκατομμύρια από όπως φαίνεται ε, έλαβε τέλος ε, το 2015 αλλά έπρεπε να ρυθμιστούν λεπτομέρειες το 2016. Λοιπόν το ερώτημα το δικό μου βάσει των ε, όσων απαντήσατε. Ωραία, αφού υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης διαφόρων περιπτώσεων και να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις στις νομοθεσίες, το πρόβλημα είναι ότι σε μια τράπεζα όπως η Deutsche Bank, που είναι συστημική τράπεζα, και ήδη απολαμβάνει εξαιρετική εύνοια διότι στην αξιολόγηση κινδύνων δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα asset τρίτου επίπεδου που εκτιμώνται ε, ε, να υπάρχουν ιστορικά στην τράπεζα. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν όπου στρεβλώνεται την τραπεζική αγορά διότι πάτε και καταδεικνύετε τον, κίνδυνο, τον πιστοτικό κίνδυνο ενώ το χρηματοπιστωτικό κίνδυνο τον ξεχνάτε τελείως. Έχετε λοιπόν αυθαίρετα λάβει και μια απόφαση να διασώσετε μια γερμανική τράπεζα, μια από τις πιο συστημικές, χρησιμοποιώντας ε, τα ε, υψηλή οικονομική, υψηλές οικονομικές δυνατότητες. Η Κασμα Μπάνκ της Ισπανίας ε, σε αυτή την περίπτωση γιατί δεν είχατε την ίδια μεταχείριση. Γιατί κάνετε τέτοια διάκριση. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά δίνεται άσχημη εικόνα σε διεθνές επίπεδο διότι προκύπτει ότι η SSM, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες ε, ε, έχουν μια σύγκρουση συμφερόντων ουσιαστικά κάνουμε αξιολογήσεις που σε καμία περίπτωση δεν είναι συγκρίσιμες με την πραγματικότητα. Για ποιο λόγο λοιπόν να πιστέψει κανείς η Τραπεζική Ένωση και σε ένα μηχανισμό, ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, όταν αυτός δεν βοηθά να αντιμετωπιστούν οι αιτίε της τραπεζικής κρίσης. Δηλαδή να πάμε να κατηγορήσουμε τις τράπεζες που υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσουν και να καταστρέψουν ε, το τραπεζικό σύστημα αλλά καταδικάζεται μόνο μερικές που δάνεισαν κάποια χρήματα στην πραγματική οικονομία και σε μικρές ε, δραστηριότητες σε μια οικονομία που είναι πιο υγιής από ότι το τραπεζικό σύστημα το οποίο περασπίζεστε εσείς. Ε, δύο λεπτά είναι η ερώτηση, λέει ο πρόεδρο. Φτάστε στην ερώτηση. Αυτό έκανα ω ερώτηση. Για ποιο το λόγο ε, δίνουμε διαφορετική μεταχείριση στη Γερμανική και στην Ισπανική τράπεζα. Γι' αυτό, αυτό ρωτάω. Uh, for your question. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ε, δεν μ' αρέσει συνήθως να αναφέρομαι σε συγκεκριμένες τράπεζες κατ' αλλά η τράπεζα που αναφέρατε εκεί δεν συνέβη τίποτα το 2015. Ήταν το 2016. Ως αποτέλεσμα η τράπεζα δεν ζήτησε τίποτα. Διότι ήταν άσχετο αυτό. Δεν ξέρω πού το βρήκατε. Δεν είναι ότι έχουμε παρόμοια περίπτωση με διαφορετικό αποτέλεσμα. Ήταν δύο περιπτώσεις εντελώς διαφορετικές. Στην πρώτη περίπτωση, στη μία περίπτωση δεν είχε τεθεί καν τέτοια απέτηση. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ποια είναι η ερώτησή σα. Ξέρω ότι το διαβάσετε στι εφημερίδε, αλλά δεν είναι επειδή βγήκε στι εφημερίδε. Ε ε, ε, ε, δεν σημαίνει επειδή βγήκε στι εφημερίδε ότι ήταν σωστό. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και θα σα συμβούλευα να επικοινωνήσετε με την ε, Ισπανική Εποπτική Αρχή και είμαι βέβαιη ότι θα σα δώσουν τι σχετικέ πληροφορίε. Τώρα, όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο για την αγορά, σε περίπτωση μη επαρκώ αποτελεσματικής εξέταση, αυτό είναι λάθος. Κατά την ολοκληρωμένη αξιολόγηση, για παράδειγμα, ήμασταν πολύ σκληροί όσον αφορά την παρεμβατική ε, αντιμετώπιση των κινδύνων της αγοράς. Και αυτό συμβαίνει διαρκώ, Διότι οι κίνδυνοι αυτοί είναι πολύ σοβαροί και του λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, ειδικότερα μετά την κρίση. Αλλά όσον αφορά εμένα και πριν την κρίση, το ίδιο έπρατα. Και πάλι εδώ, επαναλαμβάνω, αντιμετωπίζουμε ισότιμα τις τράπεζες ανάλογα με τον πιστοτικό του κίνδυνο, τον κίνδυνο για τις αγορές και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να προσθέσουμε δυσκολίες ε, που θα δημιουργηθούν από διάφορες δραστηριότητες επικίνδυνες των τραπεζών. Thank you, Barbara. Ευχαριστώ, Μπάρμπαρα Κάπελ. Äh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Νουή, είπατε τον Οκτώβριο την εξή ε, φράση. Οι τράπεζες που προσαρμόζονται θα ε, ε, ευμερίσουν, όσες δεν το κάνουν θα χρεοκοπήσουν. Δεδομένων δε των πολύ χαμηλών επιτοκίων και όλων των σκληρότερων συνθηκών ανταγωνισμού, το ερώτημα είναι πώς ακριβώς θα πρέπει να προσαρμοστούν οι τράπεζες. Μιλήσατε για το 5% απόδοση στο δεύτερο εξάμεινο αυτού του έτους, μιλήσατε για τις επενδύσεις σε υποδομές πληροφορικής και θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα ζητήματα. Το πρώτο φορό τον ανταγωνισμό και τις ρυθμίσεις, δηλαδή τράπεζες και μη τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν απαιτήσει διαφάνειας, ε, τα κριτήρια της βασιλείας κτλ. Έχουν πολύ αυστηρές ε, διατάξεις, ενώ οι σκιώδεις ε, τράπεζες εντωμεταξύ έχουν φτάσει το 1 τρίτο των χρηματαγορών ε, στην Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν, εάν θεωρείτε πως η σκιώδης ε, τραπεζική και η fintech το πρέπει, θα πρέπει στο προσεχές μέλλον να ρυθμιστούν και να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού με τις τράπεζες και αν, ε, αν έχετε συγκεκριμένες προτάσεις και χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Δεύτερη ερώτηση αφορά τον κίνδυνο κρατικών ομολόγων. Εδώ πέρα οι απαιτήσει για λόγο ομόχλευσης και τα λοιπά ε, οδηγούν τον κόσμο να επενδύει σε πιο ασφαλή προϊόντα. Όμως, για να είναι κερδοφόρες, οι τράπεζες θα πρέπει να αναμάσουν στο χαρτοφυλάκιό τους και πιο επισφαλή προϊόντα. Εσείς στο πλαίσιο αυτό λοιπόν είπατε πως δεν είναι επαναστατική προσέγγιση ή κίνδυνοι αυτοί να περιορίζονται μέσω υψηλότερων κεφαλιακών απαιτήσεων. Και σε μία ε, συνέντευξη στη Σχολή Μποκόνη στο Μιλάνο είπατε αυτό το οποίο θα ήταν επαναστατικό θα είναι να υπάρξει ένα πλαφόν στα ε, κρατικά ομόλογα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι μακροοικονομικές συνέπειες θα είχε κάτι τέτοιο για την χρηματοδότηση των κρατών και τι άποψη έχετε για το ότι θα οδηγηθούν οι τιμές προς τα πάνω εάν ταυτόχρονα γίνει και πιο δύσκολο για τις τράπεζες να εκπληρώσουν τα aero ratios. Καλέ ερωτήσει. Καλές ερωτήσεις. Ελπίζω να μην παραλείψω καμία στις απαντήσεις. Σε ό,τι αφορά την ανάγκη αναπροσαρμογής του επιχειρηματικού μοντέλου των τραπεζών ε, στις ε, τρέχουσες εξελίξεις, πρώτα απ' όλα οι τράπεζες θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές. Πάντως, ε, ο λόγος κόστος εισοδήματος είναι σχετικά υψηλός Οπότε υπάρχει δυνατότητα αύξησης αποτελεσματικότητας και μείωσης του κόστους. Σε άλλες περιστάσεις, ίσως να υπάρχει πλεονάζουσα ικανότητα των τραπεζικών, ε, της προσφοράς των τραπεζικών υπηρεσιών. Ίσως ε, είναι εκτές και κάποιες ε, συγχωνεύσεις σε κάποιες περιστάσεις, σε κάποιες χώρες για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα. Κάτι που ήδη γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Και αυτοί είναι κυρίως ε, οι τρόποι που εξετάζονται από τις τράπεζες. Δεν είναι στρατηγική βέβαια, αλλά είναι εργαλείο. Η ψηφιοποίηση βοηθάει πολύ τις τράπεζες να μειώσουν το κόστος τους και να βελτιώσουν τους δείκτες τους. Και δεν είναι ψηφιοποίηση μόνο χάρη των ε, πελατών, καλής ποιότητας ε, τεχνολογίες πληροφορίες, αυτοματοποίηση, καλή ποιότητα αυτοματοποίησης είναι ισχυρά εργαλεία που μειώνουν το κόστος λειτουργίας μιας τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό με τα μη τραπεζικά ιδρύματα και μη τραπεζικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ε, από τη στιγμή που ε, υπάρχουν ήδη κίνδυνοι, θα πρέπει να ισχύουν και οι ίδιοι κανόνες όπου είναι δυνατό στηρίζουμε πλήρω τι ε, προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπιστεί αυτή η σκιώδη τραπεζική δραστηριότητα, το shadow banking. Αν, αν κάποιοι οργανισμοί έχουν ιονή τραπεζικέ ε, δραστηριότητε ή σχεδόν τραπεζικέ δραστηριότητε, θα πρέπει να υπάγονται στου ίδιου κανόνε για να εξασφαλιστεί θεμητό ανταγωνισμό με τι υπόλοιπε τράπεζε. Και παρακολουθούμε το θέμα προσεκτικά. Επίσης, ε, χρειάζονται και οι τραπεζικές υπηρεσίες ε, για κάποιες δραστηριότητες και ίσως έτσι ε, οι τράπεζες έχουν την ευκαιρία να εξυπηρετήσουν και άλλους πελάτες. Πάντως, το θέμα του ανταγωνισμού είναι αρκετά ανοιχτό και είναι σκληρός ο ανταγωνισμός στο νέο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Και οι τράπεζες θα πρέπει να βρουν ένα καλό τρόπο και να κάνουν καλά τη δουλειά τους σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον για να επιβιώσουν. Γι' αυτό τους ζητάμε να επανεξετάσουν την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Σε ό,τι αφορά την ε, έκθεση σε ε, δημόσια, ομόλογα δημόσιο χρέους. Κάτι που το μάθαμε και από την κρίση και είναι κάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και η Τραπεζική Ένωση άλλωστε θεσπίστηκε προκειμένου να ε, αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της, ε, του δεσμού αυτής της τράπεζας με το δημόσιο χρέος, με τους ε, δημόσιους προϋπολογισμούς. Αυτή η σχέση εξετάζεται και αντιμετωπίζεται. Γι' αυτό έγινε και η Τραπεζική Ένωση. Βέβαια, είναι χρονοβόρη διαδικασία. Δεν θα ολοκληρωθεί όλη η προσπάθεια πολύ γρήγορα, αλλά καλό είναι να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό και να ξεκινήσουμε με κάτι αργό αλλά σταθερό και σταδιακό, ώστε να δώσουμε τα σωστά κίνητρα και να αποφύγουμε τις διαταράξεις ε, της ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Και ιδεοδός θα έπρεπε να ε, αποτελεί τμήμα ενός παγκόσμιου πακέτου για να μην δημιουργηθούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των ευρωπαϊκών τραπεζών. Χωσέ Μανουέλ uh, Manuel Α, σε μπέρδεψε με τον άλλο Φερνάντε. Ναι, να το γνωρίζω. Σας ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε και καλωσορίζω και την πρόεδρο του ενιαίου αποπτικού μηχανισμού, την κυρία Ντανιέλ Νουή. Έχω μια ερώτηση για την κεφαλαιοποίηση της ε, Κάισα Ζεράλτη Depositus, ε, μιας δημόσιας τράπεζας ε, ταμευτηρίου στην Πορτογαλία. Ποιος είναι ο ρόλος του, Ευρωπαϊκού του ενιαίου μηχανισμού και της ΕΚΤ σε αυτή την κεφαλαιοποίηση της Κάσιο Ζεράλ Depositus της Πορτογαλίας. Και τι ενημέρωση έγινε στην έκτη για αυτή την κεφαλαιοποίηση. Εσείς συναντηθήκατε με τον Αντώνιο Ντομίγκες, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Kaiser Herald Depositus, για να συζητήσετε και να ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης αυτής της τράπεζας. Ευχαριστώ. Η δουλειά μου ως ε, επόπτη του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού είναι να εξασφαλίσω ε, σωστή επαρκή κεφαλαιοποίηση των τραπεζών και αντιμετώπιση των αδυναμιών τους. Αυτό ισχύει και για την Kaiser Gerald Depositors που αναφέρεται, αλλά και για όλες τι ευρωπαϊκέ τράπεζε. Όταν τώρα μια τράπεζα είναι δημόσια ε, και μέτοχος κύριο είναι το κράτος, Και αυτή είναι μια κατάσταση που δεν έχει δημιουργηθεί από την κρίση μόνο, υπήρχε και από πριν, προϋπήρχε. Οπότε είναι ε, φυσιολογικό ε, η Δημόσια Τράπεζα να απευθύνεται στο ε, δημόσιο για να διεκδικεί αύξηση του κεφαλαίου. Μια και πρόκειται για Δημόσια Τράπεζα, κάτι τέτοιο γίνεται υπό τον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Η Γενική Διεύθυνση αυτή μεριμνά το δημόσιο μετοχικό κεφάλαιο που δίνεται στην τράπεζα Ε, χορηγείται υπό συνήθεις ε, προϋποθέσεις ε, παιδιτού και δεν είναι και καλυμμένες κρατικές ενισχύσεις αυτή η έχηση κεφαλαίου. Επίσης, θέλουμε η απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου να είναι αντίστοιχη με, αυτή που, με την απόδοση που περιμένουμε από ιδιωτικά κεφάλαια. Και θα σας το εξηγήσουν αυτό οι αρμόδιοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Αυτό ισχύει για όλες τις τράπεζες, όχι μόνο για τις δημόσιες. Είπατε ότι συναντήθηκα με τον κύριο Ντομίγκες όταν έγινε η αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας. Μα ακριβώς αυτό κάνουν οι επόπτες. Είμαστε επιφορτισμένη με τον σωστό και επαρκή έλεγχο και την αξιολόγηση σε διάφορα διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με το μέγεθος και τη συστημική αξία σημασία της τράπεζας. Ανάλογα με όλα αυτά, συναντούμε τους αρμοδίους της τράπεζας, τους διευθυντές ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο για μας, αυτές οι συναντήσεις και δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ιδιωτική και δημόσια τράπεζα στην περίπτωση αυτή. Η μόνη διαφορά είναι η αρμόδια γενική διεύθυνση, που είναι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, που μεριμνά οι επενδύσει ε, που κάνει το δημόσιο να είναι αντίστοιχε με τι ιδιωτικέ και να μην είναι καλυμμένε κρατικέ ενισχύσει. Ο Ιάκοπ Φον Βάιτσεκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Νουή, είναι μεγάλη μα χαρά που σα έχουμε εδώ και θα ήθελα να ξεκινήσω με το ερώτημα που σχετίζεται με το εκλογικό αποτέλεσμα σας είπα σήμερα το πρωί, το οποίο πιστεύω ότι ήταν μια επίπονη ε, υπενθύμηση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στις κυβερνήσεις και καθώς βρίσκεστε εδώ ε, στο δικό σας ε, ξέρετε εδώ στο Κοινοβουλίο έχουμε επενδύσει τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης Έχετε λοιπόν τεράστια ευθύνη πάνω σας και εμείς το γνωρίζουμε, Έχει επένδυθει, έχουν επένδυθει πολλά σε εσά. Όταν έχετε όμως μια τέτοια ευθύνη, ένα σημαντικό ερώτημα είναι τι κάνει κανείς ε, ε, ώστε να είναι αρκετά προσεκτικός. Δηλαδή πρέπει να εκαθαρίζονται οι ισολογισμοί πολύ γρήγορα, αυτό σημαίνει αυτό για σας διότι είναι υποφελές για την οικονομία και για την εμπιστοσύνη του πληθυσμού στο δικό σας ε, θεσμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να ικανοποιείτε συγκεκριμένα συμφέροντα συγκεκριμένων τραπεζών ή συγκεκριμένων κυβερνήσεων. Η αναθεωρήση ποιότητα του ενεργητικού ξεκίνησε φυσικά το 2013 και αυτό ήταν ο σκοπό τη. Και αυτό που μα λέτε σήμερα, και εγώ το υποστηρίζω έτσι ω ε, έργο, Μα λέτε ότι ακόμα δεν έχουμε task force για να επιτύχει αυτά που έπρεπε να είχαν επιτευχθεί προηγουμένως. Οπότε η ερώτηση μου προς εσάς στο πλαίσιο αυτό είναι πώς σχεδιάζετε να κινηθείτε ε, προσεκτικά μέσα στα επόμενα χρόνια και τους επόμενους μήνες ώστε να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σημαντικότατο πρόβλημα εμπιστοσύνη. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι πολύ πιο συγκεκριμένη. Αφορά το Βασιλεία 3 και 4 αν κάποιος δεχθεί ότι ε, οι κίνδυνοι ε, που σχετίζονται με τα μοντέλα είναι κάτι που θα υπάρχει ακόμη και αν βελτιώνουμε τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε τα πράγματα τότε πολύ λογικά στοιχείο μιας εποπτικής ε, στρατηγικής θα ήταν ένας δείκτης μόχλευσης τον οποίο έχουμε αλλά και πράγματα όπως ε, ε, ροές ε, αποτελεσμάτων το οποίο συζητάμε και η ερώτησή μου είναι θεωρείτε ότι είναι λογικό για να προσαρμοστούμε στη ιδιαίτερη περίπτωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Έχουμε συγκεκριμένα συμφέροντα. Πιστεύετε ότι σε ένα διεθνέ φόρουμ όπως το Βασιλεία θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα πράγματα και να επιμένουμε να μην υπάρχουν αυτές οι ροές, αλλά να βρούμε πιο έξυπνους τρόπους επίτευξη του στόχου. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, να σας πω ότι γνωρίζω βεβαίως την εμπιστοσύνη που έχει επιδείξει το πρόσωπό μου SSM είναι μια τεράστια ευθύνη και βεβαίως ε, θέλω να ανταποκριθώ σε αυτό. Όσον αφορά την συνολική αξιολόγηση με πολύ διαφανή τρόπο βρίσκουμε τις εκθέσεις οι οποίες ε, είναι μη εξυπηρετούμενες με την EBA και ζητήσαμε ένα λογικό επίπεδο προβλέψεων είτε στο λογιστικό επίπεδο που θα τα δουν οι ελεγκτές είτε ε, στο νομικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε βέβαια να πούμε ότι θα ζήσει κανείς ε, πολύ καιρό με τέτοιες ε, προβλέψεις, αλλά δεν αρκεί και να πουληθούν σε κάποιες ε, τιμές έτσι, χαμηλές για να τα ξεφορτωθεί κανείς. Τώρα περνάμε στο δεύτερο βήμα που είναι να πούμε στις τράπεζες ότι είναι καλό να έχουμε κάποιο λογικό επίπεδο προβλέψεων ε, στους ισολογισμούς, αλλά δεν επαρκεί, γιατί οι τράπεζες υπάρχουν για να χρηματοδοτούν την οικονομία, όχι για να προσπαθούν μονίμως να επιβιώσουν με βάρη που προέρχονται από την κρίση. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε επιταχύνει την διαδικασία. Είμαστε, ε, ε έτσι είναι η ζωή. Είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη την κατάσταση των διαφόρων ε, τραπεζών, τα διαφορά νομικά πλαίσια, νομικά συστήματα και όσον αφορά τα ιστορικά στοιχεία ενεργητικού από το παρελθόν αυτό το οποίο βεβαίω πρέπει να γίνει είναι μια κατά περίπτωση ανάλυση με μια όθηση των εποπτικών αρχών. Ζητάμε από τις τράπεζες να μας πούν ποια είναι τα σχέδιά τους για να αντιμετωπίσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα τις εκθέσεις, αυτές τα ανοίγματα αυτά τα οποία είναι μη εξυπηρετούμενα και ζητάμε βεβαίως περισσότερα όταν ε, θεωρούμε ότι η τράπεζα μπορεί να ανταποκριθεί. Αλλά επίσης, για το μέλλον, χάρη σε κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε δημοσιεύσει ή ίσως άλλες που θα δημοσιεύσουμε στο μέλλον, φροντίζουμε η έκθεση αυτή να αφορά μόνο στοιχεία ιστορικά, το παρελθόν και η κατάσταση αλλάζει. Για τα νέα δάνεια δεν ε, επανερχόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Όσον αφορά τη Βασιλεία, τον κίνδυνο των μοντέλων, ναι υπάρχει ένα τέτοιο κίνδυνο, αλλά εξαρτάται και από την πολυπλοκότητα των μοντέλων και τη λειτουργία. Κάποια μοντέλα δεν είναι τόσο περίπλοκα. Το λόγος μόχλευσης πράγματι είναι καλός μηχανισμός στήριξης έτσι ώστε τουλάχιστον να υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο θα προστίθεται στο λόγο μόχλευσης. Εγώ θα έλεγα ότι ε, αν κάνουμε καλή δουλειά όσον αφορά την αξιολόγηση των μοντέλων των τραπεζών και διατηρούμε την ποιότητα των μοντέλων, Ίσως να μην χρειάζεται η ροή αυτή ε, παραγωγής, αλλά αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από το επίπεδο, όπως είπαμε, της ροής αυτής. Και ένα μέρος της λύσης είναι μια ενιαία προσέγγιση που θα είναι ευαίσθητη και στους κινδύνους. Αν ε, συμβεί αυτό και νομίζω πως πηγαίνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση θα υπάρχουν λιγότερα κίνητρα για τις τράπεζες να χρησιμοποιούν μοντέλα τα οποία θα κοστίζουν ε, ε, να πιστοποιηθούν και να διατηρηθούν. Πιθανότατα δεν τα χρειάζονται ε, αν είναι απλές τράπεζες κτλ. Πολλά στοιχεία λοιπόν που κατά την απόψή μου είναι μέρος της λύσης για να έχουμε κάτι το οποίο θα είναι λογικά σταθερό και με κάποια επιμέλεια. Σας ευχαριστώ, Χωσέ Μανώλη Φερνάνδης. Θα μιλήσω γαλλικά αυτή τη φορά, για να μην χρειαστεί και διερμηνία, να με καταλάβετε απευθεία. Θεωρώ ότι η διαφάνεια είναι πάντα καλύτερη πολιτική και ο καλύτερος δρόμος. Χρειάζεται όμως και μια κουλτούρα υπευθυνότητας, γιατί μερικές φορές δεν βρίσκουμε κανέναν υπεύθυνο. Τα εθνικά κοινοβούλια δεν μπορούν να, να υποβάλουν ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Κατάλαβα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ενιαίος υποπτικός μηχανισμός δεν διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στην επανακεφαλαιοποίηση της Πορτογαλικής Τράπεζας Κάσα Γεράλντι Depositus που είναι μια δημόσια τράπεζα. Αυτή ήταν ε, η ερώτησή μου και ρώτησα πότε συναντηθήκατε με τον πρόεδρο αυτής της δημόσιας Πορτογαλικής Τράπεζας αν έγιναν επίσημα αυτές οι συναντήσεις ήταν άτυπες συναντήσεις. Ούτε και αυτό μου το απαντήσατε. Επίσης ε, ρώτησα τι είδους πληροφορίες έστειλε πήρε η ΕΚΤ για να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ε, για τις πιστώσεις, ε, για την κατάσταση της τράπεζας, για την προσωμείωση των ζημιών. Πότε έγιναν αυτές οι εκτιμήσεις και πότε στάλθηκαν αυτά τα στοιχεία. Νομίζω ότι ε, εδώ είναι η κατάλληλη ευκαιρία να επιδείξουμε διαφάνεια που όπως είπα κατά τη γνώμη μου είναι ο καλύτερος δρόμος. Ευχαριστώ και Ευχαριστώ που μιλάτε αυτά τα άψογα γαλλικά. Και έτσι με επιτρέπετε να απαντήσω και εγώ πιο εύκολα χωρίς να περάμε από τη διερμηνία. Φυσικά, καλό πράγμα η διαφάνεια, εννοείται. Υπάρχει όμως και το επαγγελματικό απόρριτο. Και ε, δεν μπορώ να δώσω με μεμονωμένες πληροφορίες για συγκεκριμένες τράπεζες. Παρ' όλα αυτά θα σας απαντήσω. Γιατί αυτό που κάνουμε για την τράπεζα αυτή είναι κάτι που κάνουμε για όλες τις τράπεζες. Δεν θα έλεγα ότι δεν είχαμε καμία ευθύνη στην επανακεφαλαιοποίηση αυτής της τράπεζας. Γιατί όταν οι τράπεζες βρίσκονται σε μία δυναμία, ε, έχουν αδυναμία είτε ως προς το κεφάλαιο είτε ως προς άλλα στοιχεία, ζητούμε από τις τράπεζες αυτές μία ανακεφαλαιοποίηση για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και τις αδυναμίες τους. Αυτό κάναμε και με τη συγκεκριμένη δημόσια τράπεζα μετά από επιτόπιους ελέγχους και διερευνητικές αποστολές. Τώρα δεν θυμάμαι απ' έξω πότε έγιναν αυτοί οι έλεγχοι και αυτές οι αποστολές. Μιλούμε όμως για μια διετία, γιατί τα τελευταία διετία αναλάβαμε τέτοια καθήκοντα. Ε, μιλούμε για το πρόσφατο παρελθόν δηλαδή. Και μετά την εποπτεία που ασκήσαμε είχαμε συζητήσεις με την τράπεζα, ε, λάβαμε τα στοιχεία, τα δεδομένα που στέλνουν τακτικά οι τράπεζες στους επόπτες, είχαμε επιτόπιους ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και έρευνα μετά από αίτημα της τράπεζας για ίδια κεφάλαια. Και αυτόματα η τράπεζα αυτή αντί να στραφεί στις αγορές για να ζητήσει χρηματοδότηση από επενδυτές, ζήτησε από τον ιδιοκτήτη της, δηλαδή το πορτογαλικό κράτος, ε, βοήθεια για την ανακεφαλαιοποίηση. Η διαφορά με τις άλλες τράπεζες που ζητούν ε, επενδύσεις από την αγορά, χρηματοδότηση από την αγορά, είναι ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υπησέρχεται εδώ για να εξακριβώσει αν τα δημόσια κονδύλια που πηγαίνουν σε τράπεζα γίνονται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Για παράδειγμα θα ρωτήσουμε ε, την τράπεζα τι απόδοση ε, έχει η επένδυση που έγινε. Θα πρέπει να είναι απόδοση αντίστοιχη με αυτή που απαιτεί αγορά για τέτοιες επενδύσεις. Αυτό εξακριβώνει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ότι ήταν αποδοτική επένδυση με όρους ιδιωτικής επένδυσης. Αλλιώς δεν δίνει η Γενική Διεύθυνση την έγκριση για την ανακεφαλαιοποίηση από το κράτος. Γιατί και άλλες δημόσιες τράπεζες, διαμερικές για παράδειγμα, πηγαίνουν στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ε, ζητώντας ανακεφαλαιοποίηση. Η ανακεφαλαιοποίηση είναι κάτι συνηθισμένο στην ιστορία μιας τράπεζας. Δεν σημαίνει ότι πρόκειται για κρατική ενίσχυση. Αν συναντήθηκα με τον κύριο Ντομίγκες, ναι, φυσικά, συναντώ όλους τους τραπέζιτες που ζητούν ραντεβού μαζί μου. Ως επόπτης ε, έχω αυτό το καθήκον. Συνάντησα λοιπόν τον κύριο Ντομίγκες, ε, ήρθε στη Φραγκφούρτη. Μάλιστα έλαβα μέρος και σε μια διάσκεψη ε, που είχε γίνει στην Πορτογαλία και μου ζήτησε να το συναντήσω. Δεν το αρνήθηκα, γιατί δεν είναι κάτι έκτακτο. Τώρα αν ήταν τυπική, επίσημη, ανεπίσημη επαφή, τι να σας πω, όταν λέω κάτι ο λόγος μου με δεσμεύει, άσχετα αν είναι τυπική ή άτυπη η ατυπη Πάντως το έργο μας ήταν το φυσιολογικό, το κανονικό έργο εποπτείας, δεν ήταν τίποτα εξαιρετικό, έκτακτο. Φροντίσαμε να είναι κατάλληλο με τις διοικητικές ε, εργασίες της τράπεζας. Ε, τα, τα, το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έγινε τίποτα κατάλληλο ή ανάρμοστο στο πλαίσιο αυτό. Ευχαριστούμε, Αλφρέτ Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρία, αξιότιμη κυρία, έχουμε καταφέρει να αποφύγουμε διπλή νομοθεσία εισάγοντα συγκεκριμένες απαιτήσει εποπτείας για συγκεκριμένες τράπεζες βασιζόμενες στην εποπτεία σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο και σε εθνικό επίπεδο με σκοπό οι κίνδυνοι να καλύπτονται ομοιόμορφα στην Ευρωζώνη. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι αντίστοιχες τράπεζες έχουν ε, τερματίσει ε, επιχειρηματικές σχέσεις με συγκεκριμένες κατηγορίες ε, ε, πελατών για διάφορους λόγους. Υπερβολικό κόστος συμμόρφωσης, κίνδυνο δραστηριοποίηση σε άλλες δικαιοδοσίες και δυσκολίες διαχείρισης κινδύνων ε, σε περίπτωση ξεπλήματος χρήματος ή ε, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αν παραμείνουν αυτά τα ζητήματα χωρίς αντιμετώπιση, μπορεί συστημικά να επηρεαστούν οι δραστηριότητες σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες με αποτέλεσμα τα προβλήματα για συγκεκριμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τράπεζες και συγκεκριμένους οργανισμούς και για ευάλωτα κομμάτια του πληθυσμού γενικότερα ο κίνδυνος μιας τέτοιας ε, επίπτωσης στο παγκόσμιο σύστημα θα απαιτήσει δράσεις πολιτικές. Αυτό θα επηρεάσει τις μικρότερες χώρες Ευρωζώνης που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Επειδή ο SSM πρέπει να διευκολύνει την συνεργασία μεταξύ τραπεζών, ποια είναι η απόψή σας για αυτό το ζήτημα και ποιες δράσεις πολιτικής θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πράγματι γνωρίζω ότι πολλές τράπεζες έχουν μειώσει σημαντικά τις ε, αντίστοιχες ε, τραπεζικές τους δραστηριότητες και αυτό μπορεί να αποτελέσει πηγή ανησυχίας για ορισμένες μικρές χώρες εντός του ενιαίου μηχανισμού υποπτίας του SSM και ε, λυπάμαι γι' αυτό αλλά δεν οφείλεται σε μένα, δεν αποτελεί απέτηση του SSM η μείωση των αντίστοιχων ε, τραπεζικών δραστηριοτήτων. Ο λόγος είναι λόγοι είναι η συμμόρφωση με συγκεκριμένους κανόνες προστασία των καταναλωτών, με κανόνες που αφορούν την καταπολέμηση του συνομοποίησης εισόδων από παράνομε δραστηριότητες. Οι απαιτήσει είναι υψηλότερε από ό,τι παλιότερα. Και έτσι οι τράπεζες έχουν μεγαλύτερη συνείδηση των κινδύνων αυτών και ως επόπτη, εγώ θεωρώ ότι καλό είναι αυτό βέβαια. Αλλά αυτή είναι η αιτία. Ελπίζω ότι με τον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό ως ενιαία δικαιοδοσία θα είναι ευκολότερο οι τράπεζες που εντάσσονται σε αυτό το μηχανισμό, στο SSM, να ε, τήρουν τις προποθέσεις. Αυτό ελπίζω πιο εύκολα. Αλλιώς δεν φαντάζομαι, δεν βλέπω να μπορώ να κάνω εγώ κάτι σε δικό μου επίπεδο. δεν δύναμε ουσιαστικά να δράσω σε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Παύλο Σάλβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ανουή που ήρθατε εδώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάποια πράγματα για το πακέτο τίτλοποίησης καθώς είμαι εισηγητής φέτος θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, όπως σας είπα, για την ιεράρχηση των διαφόρων προσεγγίσεων και δεύτερον υπάρχουν κάποιες φωνές που θα ήθελα να αυξηθεί στο Κοινοβούλιο. Η διακράτηση κινδύνου στο 20% θα ήθελα λοιπόν να μάθω την γνώμη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, ε, πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου ότι θα υπάρξει μια εφαρμογή του προηγούμενου πακέτου της Βασιλείας και αυτό από μόνο του θα δημιουργήσει σκληρότερες απαιτήσει. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Για τις απλές και διαφανείς τιτλοποιήσεις ως υποπτική αρχή πρέπει να έχουμε την κατάλληλη μεταχείριση. Δηλαδή ένα καλό προϊόν δεν χρειάζεται δώρα από τις ρυθμιστικές αρχές για να ξεκινήσει. Νομίζω πως οι προτάσεις, και αυτή ήταν η άποψη της ΕΚΤ, οι προτάσεις της Κομισιόν ήταν λογικές και εμείς τις στηρίζαμε. οι απαιτήσει ε, διακράτησης. Ε, νομίζω τώρα είμαστε στο 5%. Νομίζω λοιπόν για ε, απλή και διάφανη τηλεοποίηση. Αυτό είναι επαρκέ και λογικό. Δεν νομίζω ότι δικαιολογείται περισσότερο. Για άλλους τρόπους και άλλα είδη τίτλοποίησης, αν είναι επισφαλή, ίσως είναι μια καλή ιδέα, αλλά οπωσδήποτε κατά την απόψή μου όχι για την ε, απλή και διάφανη. Νομίζω το 5% λειτουργεί και πρέπει να διατηρηθεί για αυτού του είδους την ε, τιτλοποίηση. Ευχαριστώ κυρία Καϊλή. Thank you, uh, Mr. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την απάντησή μου, για την, για την απάντησή σας για την επιστολή μου για την Τράπεζα Αττικής που μας διαβεβαιώσατε ότι ε, θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα στο πλαίσιο του εποπτικού μηχανισμού έτσι ώστε όλες οι τράπεζες της Ευρωζώνης να έχουν υποπτία υψηλού επίπεδου και αναμένουμε βεβαίως έναν ενεργό ρόλο του εποπτικού μηχανισμού για να μην υπάρχει άνηση μεταχείριση μεταξύ του πυρήνα και της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ερώτημά μου όμως αφορά την μείωση των κόκκινων δανείων, ειδικά στις νότιες ε, χώρες, καθώς οι στόχοι του SSM και της Τράπεζας Ελλάδας δύσκολα θα επιτευχθούν δεδομένου του τωρινού νομικού και διοικητικού πλαισίου. Κάποια πρώτα βήματα έγιναν ήδη όσον αφορά κάποιες εξοδικαστικές διαδικασίες για τα εταιρικά δάνεια, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε τεράστια προβλήματα και κατά την άποψή σας έχοντας και κατά νου την έκταση της κρίσης, η επέκταση των εγγυήσεων για να προστατευτεί τουλάχιστον η κύρια κατοικία των πολιτών που βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα συζητηθεί, είναι κάτι το αποδεκτό από τον εποπτικό μηχανισμό και αν έχετε κάποιους όρους για να δεχτείτε κάτι τέτοιο ή κάποιες άλλες προτάσεις και αυτό θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, το πλαίσιο το οποίο αναφέρατε είναι περισσότερο το πλαίσιο το οποίο προέκυψε από τις ε, συνθήκες και τους όρους που είχαν θέσει τα θεσμικά όργανα στις ελληνικές τράπεζες και στην, στην κυβέρνηση της Ελλάδος. Όσο μας αφορά δεν έχουμε φτάσει ακόμα ως ε, εκεί, δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, γιατί είμαστε σε επαφές ε, και οι διαβουλεύσεις θα τελειώσουν τα μέσα Νοεμβρίου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει οι τράπεζες να εφαρμόσουν το πακέτο το οποίο θα οριστικοποιηθεί αρχές του 2017. Τούτου λεχθέντος υπάρχουν ήδη κάποιες τράπεζες οι οποίες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει και η έμφαση είναι περισσότερο συνολική όσον αφορά την έκθεση, τα ανοίγματα, τα μη εξυπηρετούμενα. Υπάρχουν διαφόρων ειδών τέτοια δάνεια ε, από επιχειρήσεις, εταιρικά μέχρι ατομικά, προσωπικά και, ακόμα και τα ατομικά μπορεί να είναι ε, φύσης επιχειρηματικής ή να αφορούν την πρωτοκατοικία όπως είπατε και τέτοια Οπότε θα δούμε τι θα μας απασχολήσει πρώτο. Φαντάζομαι ότι η πρώτη κατοικία ανθρώπων δεν θα είναι πρώτη ε, προτεραιότητα. Κατά κανόνα ξεκινάμε με επιχειρηματικά δάνεια και, ε, και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτό δεν είναι καλό μόνο για τις τράπεζες, αλλά και για τις επιχειρήσεις το να δούμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, αν θέλουν να ξαναξεκινήσουν, να λειτουργούν οι επιχειρήσεις, να έχουν νέα πίστοση από την ε, τράπεζα, πρέπει να ξεκαθαρίσουν τους ισολογισμούς τους και οι επιχειρήσεις. Οπότε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μπορούν να γίνουν εξυπηρετούμενα αν υπάρξει κατάλληλη αναδιάρθρωση. Οπότε αυτή είναι η πρώτη ε, κατεύθυνση που θα μας απασχολήσει και μετά βεβαίως ε, τα άτομα είναι πιο ευαίσθητα και δεν λέμε βεβαίως ποτέ ότι καμία τράπεζα θα έχει 0% μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Κοιτάμε τις περιπτώσεις και τον ε, μέσο όρο ταυτόχρονα του μηχανισμού που είναι γύρω στο 7% και ακόμα και τότε οι τράπεζες ε, παρουσιάζουν δικά του σχέδια για τα μη εξυπηρετούμενα, εμεί τους ρωτάμε, πιθανώ να αμφισβητούμε και υπάρχει ένα πολυετές σχέδιο μετά το οποίο καθορίζεται με συγκεκριμένα ορόσημα, αν αυτά γίνονται σεβαστά μετά η τράπεζα είναι σε καλύτερη κατάσταση, με καλύτερους όρους και βεβαίως αν ε, η τράπεζα δεν κάνει κάτι για το οποίο έχει ήδη δεσμευτεί, δεν είναι και καλή αφετηρία. Δεν έχουμε λοιπόν φτάσει ακόμα σε αυτό το βαθμό λεπτομέρειας ποιο θα είναι δηλαδή ο πρώτος ε, στόχος. Και πάλι σας λέω, οι πρώτες κατοικίες δεν είναι ο πρώτος στόχος, ε, αλλά είναι μέρος. Και και για τα φυσικά πρόσωπα ε, ίσως είναι καλή εξέλιξη να υπάρξει ένα διάρθρωση ενός ε, δανείου και να γίνει μια πίστοση η οποία θα εξυπηρετείται. Γιατί αλλιώς υπάρχει μια, ε, γιατί είναι μια βεβαιότητα η οποία φεύγει πλέον για, και για τα άτομα. Σας ευχαριστώ την κυρία Νουή. Ήταν νομίζω μια επικοδομητική ακρόαση. Η επόμενη θα είναι στις 23 Μαρτίου του 2017. Εν τω μεταξύ εμείς ετοιμάζουμε την δεύτερη έκθεση για την Τραπεζική Ένωση που επίσης θα πάει στην Ολομέλεια και θα δούμε βεβαίω και τον διάλογο με τον SSM και την κυρία Νουή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Συγχωρείτε. Ε, ε, δικό μου λάθος, λέει ο πρόεδρος. Σημείο 7. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά. Ο εισηγητής, ο κύριος Φέρμπερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Από το 1999 έχουμε μια συμφωνία με τον Καναδά για ζητήματα ανταγωνισμού την οποία επαναδιαπραγματευτήκαμε. Πρόκειται για ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των ευρωπαϊκών και των καναδικών αρχών ανταγωνισμού. Δίκαιο ανταγωνισμού μιλάμε, δεν μιλάμε για αστικέ υποθέσει ή ποινικέ υποθέσει. Έχουμε λοιπόν τις περιπτώσεις τις οποίες μια συμπεριφορά η οποία αντιβαίνει στον δίκαιο του ανταγωνισμού έχει διατλαντικές ή υπερατλαντικές συνέπειες. Η ιδέα δηλαδή βασίζεται στο ότι πλέον ε, τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να έχουν παγκόσμια διάσταση και έχουν. Και άρα θα πρέπει και οι αρχές ανταγωνισμού να μπορούν να δρουν σε παγκόσμιο επίπεδο και βεβαίως αποτελούν τέτοιες συμφωνίες μια απάντηση στην παγκοσμιοποίηση. Η συμφωνία με τον Καναδά είναι μόλις η δεύτερη τέτοια συμφωνία. Έχουμε μια με την Ελβετία σε ζητήματα συνεργασίας και εμβέας ανταλλαγής αποδεκτικού υλικού. Ο Καναδάς είναι η δεύτερη, όπως είπαμε, όλη συμφωνία και θα θυμάστε ότι στο πλαίσιο της ακρόασης κυρίας Βεστάγκερ τη συζητήσαμε να δραστηριοποιηθεί ξανά στον τομέα αυτόν και να κλείσει και άλλες τέτοιες συμφωνίες. Και βεβαίως είναι στην παράδοση των όσων είχαμε ζητήσει αυτή η συμφωνία. Προτείνω λοιπόν στην έκθεσή μου να εγκρίνουμε αυτή την συμφωνία. Γνωρίζω πως βεβαίω εδώ πέρα εμείς ε, μόνο μια σύμφωνη γνώμη θα πρέπει να εκδώσουμε και τελικά το Συμβούλιο θα αποφασίσει και πάλι καλά που μας ρωτάει την ε, άποψή μας ε, αλλά παρόλα αυτά εγώ προτείνω να συμφωνήσουμε δεν θα μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα συμφωνία γιατί είναι ακριβώς στην γραμμή των όσων έχουμε συμφωνήσει και είναι δοκιμασμένο ήδη με την Ελβετία. Πράγματα τα οποία έχουμε ήδη αναλύσει και με τα οποία έχουμε καλές εμπειρίες. Αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε κύριε Θέρβερ ε, Πρόκειται για διαδικασία συνένεσης. Άρθρο 352. Ο Άλφρετ Σάντ. Ευχαριστώ. Όπως είπε ο εισηγητής, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά για την εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού είναι καλή. Και η συνεργασία των αρχών ανταγωνισμού της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για τη διάθεση πληροφοριών ε, για να ε, παταχθούν ε, ε, δραστηριότητες που προσβάλλουν τον ανταγωνισμό είναι σωστή. Μάλιστα, η συμφωνία εξυγχρονίζει και ανανεώνει προηγούμενη με το ίδιο θέμα. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνούμε με την ε, συμφωνία αυτή, γιατί ο Καναδάς είναι χώρα που εστερνίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές ε, για θέματα ιδιωτικής σφαίρας, προστασίας δεδομένων και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι θα γίνουν σεβαστές όλες αυτές οι αρχές και από τις δύο πλευρές το, κοινο... το Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει σχετικέ διαπραγματεύσει 9 Οκτωβρίου 2008, πριν από 6, από 8 χρόνια δηλαδή. Γιατί χρειάστηκε τόσο χρόνο για να φτάσουμε στο παρόν στάδιο, Γιατί δεν υπήρχε ε, αντίθεση ω προ την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ήταν ε, διοικητική η φύση των συμφωνιών και όλοι συμφωνούσαν στην ανάγκη πρόοδου. Έπρεπε να είχαμε προχωρήσει πολύ γρήγορα. Μήπως χάνω κάτι. Μήπω υπήρχαν ε, ε κρυφές ε, ανησυχίες ή προβλήματα. Τελικά ε, ε, υλοποιήθηκε η συμφωνία παράλληλα και άσχετα με τη ΣΕΤΑ. Πώς είναι δυνατόν όμως να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συζήτηση ως ευκαιρία για τη συζήτηση για το ΣΕΤΑ, γιατί και η ΣΕΤΑ έχει ένα κεφάλαιο για την κοινή υλοποίηση πολιτικών και διαδικασιών που καταπολεμούν ε, πρακτικές κατά του ανταγωνισμού. Αναφέρονται στο άρθρο 17.2 και τα μέτρα για να παταχθούν τέτοιε ε, συμπεριφορέ βάρο του ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι διαφανή, να μην συνιστούν διακριτική μεταχείριση και να είναι δίκαια. Και οποιαδήποτε ε, εξαίρεση από το δίκαιο ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι διαφανή. Και επίση θα πρέπει να δημοσιεύονται τέτοιε εξαιρέσει με βάση τι αρχέ ανταγωνισμού των συμβαλωμένων μερών. Οπότε η υπογραφή της συμφωνίας και η κύρωση συνάδουν πλήρως και με τη συμφωνία ΣΕΤΑ. Πάντως η παρούσα συμφωνία ε, ε, που είναι τεχνική, αν είχε ολοκληρωθεί, καλό θα ήταν να είχε ενταχθεί στην ίδια τη ΣΕΤΑ από το να ε, δρομολογείται ξεχωριστά και παράλληλα. Η κόρα Βανίδερ Χόιντεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την έκθεση, τον κύριο Φέρμπερ. Θα είμαι σύντομη. Πιστεύω ότι η πρόταση αυτή αποτελεί μια θετική εξέλιξη για την παγκόσμια οικονομία. Σε μια πραγματικά ελεύθερη αγορά δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε από εθνικές δικαιοδοσίες και σύνορα για τι υποθέσει ανταγωνισμού. Οι πιο ανταγωνιστικέ αγορέ θα δώσουν όθηση στην ανάπτυξη και στι επενδύσει, κάτι που χρειαζόμαστε. Εν ώψη του ΣΕΤΑ, αποτελεί ένα βήμα προ τη στενότερη συνεργασία, τι ανοιχτέ αγορέ και την καλύτερη προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις παραβίασης, ε, οι περιπτώσεις παραβίασης του δικαίου θα ανοιχνεύονται καλύτερα και αυτό είναι προτιμότερο για τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Καλωσορίζω την προστασία των δεδομένων που έχει συμπεριληφθεί στη συμφωνία. Ένα στοιχείο ακόμα μου δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Η πρόταση δεν εισάγει καμία υποχρέωση αλλά αφήνει περιθώριο διακριτική μεταχείριση όσων, διακριτική ευχέρειας, συγγνώμη, όσον αφορά τα σημαντικά συμφέροντα. Αυτό το σημαντικά, τι συμφέροντα εννοούμε, πώς αυτά θα καθορίζονται και από ποιον. Είναι πολύ ασαφής αυτή η περιγραφή, πιστεύω. Αλλά αυτό είναι το μόνο ερωτηματικό που έχω όσον αφορά την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Για την ΚΟΕ, Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μας, η GUNGL, ε, αντιτάσσεται στην διαφορετική λειτουργία της πολιτικής ανταγωνισμού. Γιατί είναι σαφές ε, τι συμφέρονται εξυπηρετεί. Τα ευρωπαϊκά ολιγοπόλη είναι όλο και μεγαλύτερα. Ένα σημαντικό αριθμό δημοσίων εταιριών και δημοσίων τομέων έπεσαν σε ιδιωτικά χέρια ή μετατράπηκαν ε, με βάση τις ε, αρχές ανταγωνισμού. Ε, άνθρακας, αυτοκινητοβιομηχανία, ταμιευτήρια, χαλιβουργία. Η πολιτική ανταγωνισμού ποτέ δεν ήταν πραγματικό μηχανισμό προστασία των συμφερόντων καταναλωτή. Το αντίθετο, εξυπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών. Και μάλιστα η παρούσα Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά για τον ανταγωνισμό ελάχιστα προσθέτει κατά τη γνώμη μας ό,τι αφορά την ενημέρωση ή τη συνεργασία για την καταπολέμηση των μεγάλων ιδιωτικών ολιγοπολίων και κρατά την αδιαφάνεια και τη διακριτική ε, ευχέρεια στη λειτουργία των αρχών ανταγωνισμού. Μήπω είναι τυχαίο που η αναθεώρηση αυτή τη συμφωνία με τον Καναδά συμπίπτει με τη συμφωνία ΣΕΤΑ που θα ενισχύσει την ε, συνεργασία ιδιωτικών ολιγοπολίων με τι αρχέ ανταγωνισμού και θα ανοίξει ακόμη περισσότερο τι δημόσιε υπηρεσίε ε, στο ιδιωτικό κεφάλαιο και από τι διώχθε του Ατλαντικού. Δεν είναι τυχαίο κατά τη γνώμη μα, γιατί το αντίθετο, η συμφωνία αυτή ενισχύει τέτοιε συνέργειε και αναφυσβήτητα ενισχύεται και η δική μας αντίσταση στη συμφωνία αυτή. Ευχαριστούμε. Μπορούμε να ξαναδώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, όχι, το ΙΕΝΕΦ e έχει κάποιον ομιλητή, δεν με ενημέρωσαν. Ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Πάντα το ΙΕΝΕΦ e λέει ο εισηγητής. Α, μου επιτρέπετε, εντάξει. Η Συμφωνία για τη Στενότερη Συνεργασία αυτή είναι από το 1999, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αποτελεσματική για τέτοιες ε, διατλαντικές διαδικασίες. Ελπίζω η νέα συμφωνία με την Ελβετία να αποτελέσει καλό υπόδειγμα για τη συμφωνία με τον Καναδά και οπωσδήποτε είναι αναγκαίο η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος ε, θα ταιριάζει για το διεθνές εμπόριο του 2016 και των επομένων ετών. Δύο τρίτα νομίζω των αποφάσεων ε, ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούσαν τρίτες ε, χώρες και 78% αφορούσαν επίσης οι αποφάσεις για καρτέλ ε, με τρίτες χώρες, οπότε έχουν μεγάλη σημασία οι τρίτες χώρες ε, όταν μιλάμε για τέτοιες συμφωνίες. Ε? Ο εισηγητής λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, εδώ μιλάμε για το δίκαιο του ανταγωνισμού, όχι για τη ΣΕΤΑ. Να το πω αυτό. Δεν έχει ούτε μία σχέση με τη ΣΕΤΑ. Είναι άλλη συμφωνία. Και δεύτερον, οπωσδήποτε να γίνει μια συζήτηση αρχών για το δίκαιο του ανταγωνισμού, αλλά να παρατηρήσω επίσης επί της αρχής ότι το θέμα της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και των υπηρεσιών δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό που παρέχουν τις υπηρεσίες και είναι μόνο περιφερειακό όσον αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού. Οπότε δεν θεωρώ πως η συμφωνία με τον Καναδά είναι η στιγμή για να γίνει μια συζήτηση αρχών για το δίκαιο του ανταγωνισμού. Ε, οπωσδήποτε, ε, συνάδελφος βεβαίω είναι ευπρόσδεκτη στην υποεπιτροπή μας για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Αλλά η παράκλησή μου είναι να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο πάντα λέγαμε στην Κομισιόν ως Κοινοβουλιοχώρα για τη δικιά σου ερώτηση. Ευχαριστώ να δώσω εξηγήσεις, αλλά... Όπως λες, δεν ξέρω τώρα ποιες είναι οι σημαντικές ε, διαδικασίες ε, τις οποίες αναφέρεις. Έχουμε, εν πάση περιπτώσει, καιρό για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί, ε, όπως σας είπα, μας επέτρεψε το κοινοβούλιο να εκφέρουμε άποψη, οπότε ελπίζω κόρα να μπορέσει να απαντηθεί και η δικιά σου ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τελειώνει αυτό το σημείο. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται απλά για μια σύμφωνη γνώμη, οπότε θα επανέλθουμε στο χρονοδιάγραμμα της ψηφοφορίας. Τελειώνουμε με αυτό το θέμα λοιπόν και περνάμε στο επόμενο να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο των Πρόσκης. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκη ε, σε αυτό το διαρθρωμένο διάλογο, ο οποίος είναι και ο πρώτος ε, με τον Αντιπρόεδρο από τότε που ανέλαβε το χαρτοφυλακείο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συγγνώμη. Οπότε καλωσορίζουμε αυτή την ευκαιρία για μια ανταλλαγή απόψεων για πολλά σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον τομέα αυτό Αναμένουμε το νέο πακέτο CRD, θα έχουμε το πρώτες ψηφίσματος CCP και φυσικά και την Τραπεζική Ένωση και την Κεφαλή Αγορών συμπεριλαμβανομένων των εργασιών για την τιτλοποίηση. Από ό,τι καταλάβαμε σήμερα έγινε και μια συζήτηση για την PRIPS. Έχουμε τεράστια θεματολόγιο και είναι πολύ καλό που έχουμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα αυτά μαζί σας. Και δίνω λοιπόν το λόγο στον Αντιπρόεδρο κύριο Ντομπρόφσκη, ο οποίο πρέπει να αναχωρήσει τι 6.30 από ό,τι κατάλαβα, οπότε θα είμαστε πολύ αυστηροί με τη διαχείριση του χρόνου. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Uh, thank you, uh, Mr. President, honorable members of... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση αυτή και για την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Φυσικά σήμερα είναι μια ειδική ημέρα, χαρακτηρίζεται από το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών και πιστεύω ότι καλό είναι να συζητήσουμε πώς θα ενισχύσουμε το χρηματοπιστωτικό μας τομέα, πώς θα το διατηρήσουμε σταθερό, θα υποστηρίξουμε τις επενδύσεις και την αηφόρο ανάπτυξη στην Ευρώπη. Οι εργασίες μας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εντάσσονται σε μια ευρύτερη μακροοικονομική στρατηγική ε, βάσει της σημερινής ε, αβεβαιότητας και θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σημαντικό να παραμένουμε προσπελμένοι σε αυτό που κάνουμε, να συνεχίσουμε με τις ε, οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές, με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες και να βεβαιωθούμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Η προσέγγιση μας αυτή θα περιγράφεται στην ετήσια έκθεση της ανάπτυξης ε, που πρόκειται να εκδοθεί. Όσον αφορά την ευρύτερη οικονομική κατάσταση, παρατηρούμε ότι οι οικονομίες μας ε, παραμένουν ανθεκτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ανάπτυξη σε όλα τα κράτη-μέλη του χρόνου. Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν. Σχετίζονται με το υψηλό επίπεδο βεβαιότητας και εμεί ω υπευθύνοι χαράξη πολιτική πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη αυτή και να παράσχουμε βεβαιότητα όπου μπορούμε. Αυτό ισχύει και για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Εδώ χρειάζεται να προβούμε σε σημαντικέ μεταρρυθμίσει που συμφωνήθηκαν τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα, για την πρόθεση νέων πηγών επένδυση, εμβαθύνοντα τι κεφαλαγορέ τη Ευρώπη και χτίζοντα την Ένωση αγορών. Θα συζητήσουμε λοιπόν πώ μπορούν να γίνουν όλα αυτά μαζί σήμερα. Α ξεκινήσουμε με τις κεφαλαίες Με την Ένωση Κεφαλαίων Αγορών το Σεπτέμβριο δημοσιεύσαμε μια ανακοίνωση που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μα ε, να εφαρμόσουμε το σχέδιο δράση του 2015, να επιταχύνουμε και να είμαστε πιο τολμηροί όπου μπορούμε. Και είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ αυτό το έργο. Να διατηρήσουμε την ορμή και να δείξουμε ότι η Ευρώπη παίρνει στα σοβαρά την ε, εμβάθυνση των κεφαλαίων και βασίζεται σε εσά ε, για τα πρώτη σειρά μέτρων. Έχω στο νόμο μου τις προτάσεις ανακαίνησης του σημερινού καθεστώτος και να διευκολύνουμε ε, την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου ε, στι κεφαλαιογορέ από τι επιχειρήσει. Η πρότασή μα να ξεκινήσουμε τι αγορέ τυκλοποίηση, καθορίζοντα απλέ ε, διαφανεί τυκλοποιήσει, τυποποιημένε, βάσει των εργασιών ανεξαρτήτων οργανισμών τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η πρότασή μα ενίσχυση των αγορών τη Ευρώπη και υποστήριξη των κοινωνικών επενδύσεων, τροποποιώντα τι νομοθεσίε που διέπουν τα ευρωπαϊκά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και ε, τι κοινωνικέ επιχειρήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές ε, Πίτρ Γέζεκ, Πολτάν, Παμπλο Ζάλμπα και Σύρπα κάναν ε, στις προσπάθειές τους να γεφυρώσουν τις διαφορές και να επιτύχουν συμφωνίες. Οι προτάσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να υποστηριχθούν οι επενδύσεις με αυξή της χρηματοδότησης προς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ανάκαμψης στην Ευρώπη. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν, ας δώσουμε απτά αποτελέσματα και ας προχωρήσουμε στην άρση ορισμένων ε, παλιών εμποδίων στην ελεύθερη ε, κίνηση κεφαλαίων στην Ευρώπη. Να αναφέρω τρία από αυτά. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να εξετάσουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις ε, ως προς την αφαιρεγγιότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια πρόταση τις επόμενες εβδομάδες για την υποστήριξη της αποτελεσματική αναδιαρθρώσης βιώσιμου χρέου επιχειρήσεων ώστε να δίνεται μια δεύτερη ε, ευκαιρία στις επιχειρήσεις και θα δούμε τα διάφορα καθεστώτα για να δούμε ποια λειτουργούν σωστά. Δεύτερον, ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα φορολογικά καθεστώτα και αλληλεπιδρούν σε ολόκληρη την Ευρώπη ε, μπορεί να αποτελέσει φραγμό προ τι επενδύσει, Οπότε θέλουμε να αναπτύξουμε ένα κώδικα διοντολογία για να προωθήσουμε τι βέλτιστες πρακτικέ. Ε, ε, όσον αφορά το χειρισμό του φόρου παρακράτησης και επίσης έχουμε παρουσιάσει ε, προτάσεις ε, στο πλαίσιο της ενιαίας εταιρικής φορολογικής βάσης, ενοποιημένης φορολογικής βάσης των εταιριών για να μειώσουμε το στρέβλωση υπέρ του χρέου στα φορολογικά μα συστήματα. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μια ενιαία αγορά για τι ατομικέ συντάξει. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύτιμο συμπληρώμα για τι κρατικέ και τι εργασιακέ συντάξει ε, συζητάμε για το πώς θα δημιουργήσουμε ένα σχετικό πλαίσιο. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις και τώρα ε, μελετάμε την διατύπωση των απαντήσεων και βλέπουμε κατά πόσο θα χρειαστεί να νομοθετήσουμε του χρόνου. Επίσης θέλουμε να υποστηρίξουμε τη βιώσιμη ε, βιώσιμα οικονομικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να δαπανίσει τουλάχιστον 20% του προπολογισμού από το 2014 στο 2020 για την κλιματική δράση και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαθέσουμε περισσότερα πράσινα ταμεία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Αλλά οι προσπάθειε αυτέ θα πρέπει να πάνε πέρα από τα δημόσια οικονομικά. Με όλα αυτά υπόψη, η Κομισιόν να δημιουργεί μια ομάδα εμπειρογνωμών υψηλού επίπεδου για να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βιώσιμα οικονομικά. Εξετάζουμε τι εξελίξει ε, στην αγορά των πράσινων φορολόγων και τι δυνατότητε χρηματοδότηση επενδύσεων αποτελεσματικών ω προ του πόρου. Για να αυξήσουμε τη διαφάνεια για τι εταιρείε, έχουμε συμφωνήσει την οδηγία για την μη οικονομική υποβολή εκθέσεων που θα μεταφερθεί μέχρι τα τέλη του έτου. Η πρόσφατη συμφωνία για τη ε, θεσμική και εργασιακή συνταξιοδότηση του Brian Hayes εδώ στο Κοινοβούλιο θα ενθαρρύνει τα, να λαμβάνονται υπερβολικοί παράγοντε στι επενδυτικέ αποφάσει και η Κομισιόν έχει ξεκινήσει μια δημόσια ε, διαβούλευση για τι μακροχρόνιε και βιώσιμε επενδύσει και τι προκλήσει που έχουν να αντιμετωπίσουν οι θεσμικοί επενδυτέ σε αυτόν τον τομέα. Η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών θα πρέπει να παράσχει αποτελέσματα και για τους λιανικούς επενδυτές. Οι δράσει μας μετά από την πράσινη βίβλο θα εστιαστούν στην άρση των εμποδίων ε, όσον αφορά την αγορά οικονομικών υπηρεσιών από καταναλωτές, ε, των σωστών ε, ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπου και να βρίσκονται στην Ευρώπη, θα διευκολύνουν τη σύγκριση των προϊόντων και θα διασφαλίζουν ότι οι μηχανισμοί θα λειτουργούν σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Θα υπάρχει υποστήριξη προ τι επιχειρήσει που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίε διασυνοριακά και θα διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη εκμεταλλεύεται στο έπακρο το fintech και την τεχνολογική καινοτομία για όλα αυτά, διατηρώντα ταυτόχρονα την ισχυρή προστασία των καταναλωτών. Εδώ είμαστε ευγνώμονε για την έκθεση του Ολελούντβιξον στον τομέα και θα παρουσιάσουμε ένα σύνολο δράσεων μετά το νέο έτος. Τώρα επιτρέψτε μου να περάσω στον τραπεζικό τομέα. Ε, λαμβάνοντα δράση για την εμβάθυνση των κεφαλαίων αγορών μα, συνεχίζουμε τι εργασίε ενίσχυση του πλαισίου για τον τραπεζικό τομέα τη Ευρώπη. Ο ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα είναι πολύ ισχυρότερο και έχει κεφαλαιοποιηθεί καλύτερα από ό,τι πριν ε, την κρίση. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τα πρόσφατα stress test, αλλά παραμένουν κάποιε δυσκολίε. Πολλέ τράπεζε δυσκολεύονται να δώσουν πιστώσει στην οικονομία τη Ευρώπη σε ένα περιβάλλον χαμηλή ανάπτυξη, χαμηλού πληθωρισμού και χαμηλών επιτοκίων. Οι τεχνολογικέ εξελίξει δημιουργούν νέε ευκαιρίε αλλά και προκλήσει προκλήσεις ε, για τα καθιερωμένα επιχειρηματικά μοντέλα. Το να βρούμε τις σωστές απαντήσεις ε, θα το καταφέρουμε με τη βοήθεια του τραπεζικού τομέα. Αλλά προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Κομισιόν είναι να παράσχει το σωστό περιβάλλον για να γίνονται όλα αυτά ασφαλώ και αποτελεσματικά. Θέλουμε να ενισχύσουμε την Τραπεζική Ένωση με τη δική μα πρόταση για ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό ασφάλιση των καταθέσεων. Οπότε χαιρόμαστε που προχωρούν τώρα αυτέ οι εργασίε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που συζητάτε το σχέδιο έκθεση τη Έστερ Ντελάγκε. Για να αντιμετωπιστούν τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων, τώρα παρέχουμε τεχνική υποστήριξη μέσω τη υπηρεσία μα υποστηρίξει διαρθρωτική μεταρρύθμιση και διατηρούμε την πίεση Στι συγκεκριμένε ε, συστάσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε έξι κράτη-μέλη και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να βρούμε λύσει ε, βάσει των υπαρχών των κανόνων ε, εξηγήσεω των τραπεζών και κρατική ενίσχυσης. Αργότερα το μήνα αυτό η Κομισιόν θα υιοθετήσει μια πρόταση τροποποίηση του κανονισμού και τη οδηγίας κεφαλαιακών απαιτήσεων η οποία θα αντιμετωπίσει δύο μέτωπα. Πρώτον, του κινδύνου που απομένουν στον τραπεζικό τομέα με την υλοποίηση των διεθνών προτύπων που έχουν συμφωνηθεί από την Επιτροπή τη Βασιλεία και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα με τρόπο που να υποφελούν ε, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δανείζουν στην ευρύτερη οικονομία. Δεύτερον, να θεωρούμε την νομοθεσία μας ώστε να γίνει πιο αναλογική. Έτσι προωθούμε την νομοθεσία μας ε, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο φιλική προς την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό κάναμε έκκληση για αποδεικτικά στοιχεία και βασιζόμαστε και στις εργασίες του Κοινοβουλίου αυτού και στην εκθέση του Μπουρκαντ Μπάλτ πιο συγκεκριμένα και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την έκκληση για όλε τι νομοθεσίε που αφορούν χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο προσαρμόσεων προσαρμογών για την αύξηση τη χρηματοδότηση στην ευρύτερη οικονομία και να κάνουν, θα στήσουμε την νομοθεσία πιο αναλογική παρέχοντα του ίδιου στόχου. Να δούμε κατά πόσο το βάρο τη συμμόρφωση μπορεί να μειωθεί για τι επιχειρώσει και κατά πόσο οι κανόνε μα μπορούν να γίνουν πιο συνεκτικοί και πιο προορατική. Θα χρησιμοποιήσουμε τι αναθεωρήσει του κανονισμού κεφαλαίων απαιτήσεων και του κανονισμού υποδομών Ευρωπαϊκή Αγορά για να προτείνουμε κάποιε άμεσε αλλαγέ. Συνεχίζουμε επίση να εξετάζουμε του άλλου πηγού κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ελπίζουμε να επιτευχθεί μια συμφωνία για τα ε, ταμεία των χρηματαγορών μέχρι τα τέλη του έτου και να επιτευχθεί μια κάποια ισορροπία μεταξύ του μετριασμού των κινδύνων στι αγορέ, στι χρηματαγορέ ενώ να διατηρούνται ως ένα βιώσιμο προϊόν ε, που να καλύπτει τι ανάγκε των επενδυτών. Χαιρόμαστε για τι εργασίε τη Νίνα Γκίλ στον τομέα αυτό. Πριν τα τέλη του έτου θα κάνουμε μια πρόταση για την ε, ε Central Party Recovery and Resolution. Η πρότασή μα θα βασιστεί στου υπάρχοντε ευρωπαϊκού κανόνε, ειδικότερα στον κανονισμό ε, υποδομών ευρωπαϊκών αγορών και στην οδηγία ανάκαμψης και εξηγιασής των τραπεζών. Θέλουμε να δείξουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη συνοχή στην νομοθεσία αυτή και να τα αποκριθούμε στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των CCP ώστε να είμαστε απολύτως έτοιμοι σε περίπτωση που κάτι πάει λάθος του χρόνου θα ε, παρουσιάσουμε προτάσεις επικαιροποίησης του μακροπροληπτικού μας πλαισίου. Ε, οι διαβουλεύσει μα έχουν μόλι τελειώσει, μελετάμε τι απαντήσει και ζυγίζουμε τα επιχειρήματα ώστε να φτιάξουμε ένα ισχυρότερο μακροπροληπτικό πλαίσιο με πιο αναλογικού κανόνε και με πιο αποτελεσματικού θεσμού όπω η ESRB. Να αναφέρω στα σύντομα τον τη κανονισμό PRIPS όπου εξέφρασε δυσαρέσκεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο PRIPS. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι νομοθεσία για του καταναλωτέ και η πρώτη μα υποχρέωση σε όλη τη διαδικασία είναι προς τον καταναλωτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αξιολογήσει προσεκτικά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματο. Εμεί συνεργαζόμαστε με, την Ευρωπαϊκή, ε, με τις ευρωπαϊκές Επιπτωτικέ αρχές για να εξετάσουμε τις ανησυχίες και θα στείλουμε σήμερα την ε, τι προτάσει μα έτσι. Το RTS θα προταθεί εκ νέου χωρί περαιτέρω καθυστερήσεις. Και σήμερα η Κομισιόν έχει επίση προτείνει μια παράταση 12 άμυνη για τον κανονισμό πριν ώστε οι εταιρείε να έχουν χρόνο να προετοιμαστούν για του νέου κανονισμού που θα τεθούν σε ισχύ και να υπάρξει χρόνο οριστικόποίηση του αναθεωρημένου RTS. Όλα αυτά γίνονται βάσει κοινή κατανόηση, ότι ότι δεν πρόκειται να ξανανοίξουμε την ομοθεσία επίπεδου 1. Ε, συμπερασματικά, κυρίε και κύριοι, αυτό είναι απλά ένα δείγμα των εργασιών μας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και όπως βλέπετε συνεργαζόμαστε για να βρούμε τη σωστή ισορροπία για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση προς την οικονομία προστατεύοντας τους καταναλωτές και να διατηρήσουμε το χρηματοπιστωτικό μας τομέα ανταγωνιστικό και δυναμικό αλλά ασφαλή. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας ώστε να προωθήσουμε αυτό το θεματολόγιο μέσα στι επόμενε εβδομάδες και μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Vice Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Συμφωνούμε πάρα πολύ με το πρόγραμμα αυτό και επιβεβαιώνω ότι συμφωνούμε ακριβώ στο να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία και όχι μόνο η νομοθεσία επίπεδου 1. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα με τις παρεμβάσεις μας. Πρώτος ο αντιπρόεδρος μας, ο κύριος Ζάλμπα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω ισπανικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα, να σας ενημερώσω ότι έχετε αναλάβει ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο και από αυτά τα οποία είπατε είναι σαφές ότι είστε πολύ αποτελεσματικός και σας συγχαίρω. Η εκθέσεις ε, τις οποίες αναφέρατε οπωσδήποτε είναι σημαντικές και είμαστε οπωσδήποτε διατεθειμένοι αλλά θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάτι άλλο ξέρω ότι συναντηθήκατε με Ισπανούς και Πορτογάλους υπουργού στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου θα έλεγα πως ε, υπάρχει μια σχεδόν ομόφωνα θετική απόφαση, ε, άποψη για τις αποφάσεις που έλαβαν οι δύο χώρες και επίσης ομόφωνη συμφωνία του Κοινοβουλίου για να πούμε ότι είμαστε κατά του παγώματος ε, των κονδυλίων. Ήθελα μια αξιολόγηση αυτής της ακρόασης στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου που έγινε χθε ε, στην Αρμόδια Επιτροπή. Ναι, σίγουρα. Αυτό το θέμα κάπως ξεφεύγει από τον διαρθρωμένο διάλογο χθες καταλήξαμε σε μια κοινή θέση. Ε, μπορείτε πάντως να το σχολιάσετε αν θέλετε. Για το διαφρομένο διάλογο. Φυσικά. Έχουμε επίγνωση της έκβασης του διαρθρωμένου διαλόγου και της έκκλησης να μην ε, διακοπούν τα κονδύλια, να μην γίνει αναστολή των κονδύλιων προς την Ισπανία και Πορτογαλία. Αυτό θα το λάβουμε υπόψη κατά την εκπόνηση του πακέτου αποφάσεων. Εμείς θέλουμε να εκπονήσουμε ένα πακέτο αποφάσεων και τις, α, ε, τα, σχέδια, τα δημοσιονομικά σχέδια στις 16 ε, Νοεμβρίου που θα εξελογήσουμε τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τον κανονισμό Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στις ιδιαίτερε περιπτώσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας θα εξετάσουμε τη συμμόρφωση και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου στα πλαίσια της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Μέχρι πρόσφατα πάντως δεν είχαμε ε, κανονικές κυβερνήσεις, αλλά υπηρεσιακή, υπηρεσιακή κυβέρνηση στην Ισπανία για πολύ καιρό. Και το σχέδιο προϋπολογισμού υπευλήθη με βάση ένα σενάριο σχεδόν μηδενικών αλλαγών. Πάντως είχαμε ήδη λάβει την επιστολή από την Ισπανία, από τον ε, Υπηρεσιακό Υπουργό Οικονομικών, τον Λουίς Δεγκίντες, με την δέσμευση της κυβέρνησης ε, να τηρήσει την απόφαση του Συμβουλίου και τη δημοσιονομική προσωμείωση που περίεχε. Και αυτό μας καθησυχάζει και θα το λάβουμε υπόψη κατά την απόφαση αναστολής ή όχι των κονδύλιων προς την Ισπανία. Όλους αυτούς τους ε, παράγοντες θα τους λάβουμε υπόψη, αλλά δεν μπορώ να προεξοφλήσω την απόφαση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα. Πάντως, σίγουρα αφού γραζόμαστε τα μηνύματα που στέλνετε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώ το εκτιμούμε ιδιαίτερα, λέει ο πρόεδρο, ο Πέτερ Ζήμων. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω. Η μία αφορά τις τιτλοποιήσεις, η άλλη αφορά το σύστημα καταθέσεων. Στις τιτλοποιήσεις συζητάμε αυτή τη στιγμή πόσον κίνδυνο θα διακρατήσει αυτός ο οποίος θα εκδώσει τους τίτλους για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε τις ίδιες λανθασμένες εξελίξεις που είχαμε στην οικονομική κρίση και στη ΣΥΠΑ. Εδώ πέρα συζητάνε και στην ομάδα μου ότι θα πρέπει να διακρατηθεί μέχρι και 20%. Άλλοι ήθελαν, θα ήθελαν ένα 5%. Θεωρείτε πως θα μπορούσαμε να διαφοροποιούμε ανάλογα με το τι τιτλοποιείται. Γιατί προτείνω μια τέτοια διαφοροποίηση. Στον τομέα του τι τιτλοποιείται έχουμε πολλές διαφορές στην Ευρώπη. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, στα στεγαστικά, τιτλοποιήσεις μάλλον στεγαστικών, ένα ποσοστό μη εξυπηρετούμενων που είναι τριπλάσιο από ό,τι τα δάνεια για αυτοκίνητα. Θεωρείτε λοιπόν πως θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση ανάλογα με το αντικείμενο της τιτλοποίησης του ε, ποσοστού διακράτησης κινδύνου. Ερώτηση πρώτη. Ερώτηση δεύτερη αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Μιλήσατε για τις επιχειρήσεις ε, και τις διαδικασίες ε, χρεοκοπίας. Και η κυρία Ντελάγκη μίλησε για τη διαδικασία μετάβασης από μία φάση ασφάλισης σε μία φάση πλήρους κινητικοποίησης από τη φάση 2 στη φάση 3 και είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο πτωχευτικό δικαίωμα στην Ευρώπη. Αν λοιπόν δούμε το θέμα αυτό ε, του πτωχευτικού δικαίου θα καλύψετε και αυτόν τον τομέα. Κάτι δηλαδή ανάλογο με αυτό το οποίο πρότεινε η κυρία Ντελάγγεν στην έκθεσή της για το έντις. Σας ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις υπήρχαν. Πρώτη για την τιτλοποίηση και τη διακράτηση του κινδύνου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, αλλά βασικά η δική μας πρόταση ε, διατηρεί την υφιστάμενη προσέγγιση στην διακράτηση του κινδύνου και φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά, των ρυθμιστικών αρχών, των κεντρικών τραπεζών, των Υπουργείων Οικονομικών, πώς λειτουργούν επαρκώς ε, αυτή τη στιγμή αυτά. Ε, δεν υπάρχει κάποιο άλλο νούμερο στο οποίο υπάρχει τόσο μεγάλη συμφωνία από διαφορετικούς συμμετέχοντες και η Επιτροπή των Ευρωπαίων Τραπεζικών εποπτών, ε, προκάτοχος της EBA, είχε πει το 2009 ότι δεν μπορεί να βρει στοιχεία ότι η αλλαγή, η αύξηση του ποσοστού διακράτησης ε, από το 5% θα ε, είχε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη διαφόρων ανεπιθύμητων συνεπειών. Και μια παρόμοια προσέγγιση βεβαίως είχε και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή το τέλος του 2014 όταν είχε γράψει την σχετική της έκθεση για την δεύτερη επιμέλεια, την τιτλοποίηση και είχε πει πως οι υφιστάμενοι κανόνες διακράτησης του κινδύνου αντιμετωπίζουν έναν το κίνδυνο και λειτουργούν επαρκώς. Οπότε οι ρυθμιστικές αρχές λένε πως το υφιστάμενο σύστημα φαίνεται ότι έχει αποτελέσματα. Αυτή είναι η βάση της πρότασής μας. Βεβαίως, αναμένουμε την απόφαση του Κοινοβουλίου και είμαστε έτοιμοι να έχουμε μια συζήτηση ανοιχτή και επικοδομητική για να βρεθεί μια λύση. Για να εξηγήσω δηλαδή πώς, γιατί η πρόταση της Κομισιόν έχει όσο έχει μετά για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Αυτή τη στιγμή μια που το σχέδιο έκθεσης ε, μόλις πρόσφατα έγινε διαθέσιμο Πρέπει να αξιολογήσουμε την έκθεση ακόμα. Ξέρουμε ότι δεν έχει ψηφιστεί ούτε στην Επιτροπή ακόμα. Πριν καταλήξουμε λοιπόν σε κάποια συμπεράσματα και σε σχόλια. Γενικά θα έλεγα ότι από την πλευρά της Κομισιόν τονίζουμε ότι η μείωση του κινδύνου πρέπει να πάει χέρι-χέρι με την με το να τον μοιραστούμε από κοινού. Σας ευχαριστώ και βέβαια πρέπει να είναι και κάτι το οποίο θα στέκει νομικά. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν και άλλα που δεν μπορούν να γίνουν σε έναν κανονισμό. Λοιπόν, και η Σουινμπορν. Ευχαριστώ. Μόλις α, ε, αυτές από μια διάσκεψη για τις, α, ε, ευρωπαϊκή διάσκεψη για τις ε, συντάξεις, Πέρσι είναι πρώτη διαβουλεύσει ε, για την ε, αξιολόγηση και την αναθεώρηση του συστήματο και έκτοτε εξετάζεται ε, κάποιε αλλαγέ. Στο ΕΜΗΡ έχουμε κάποιε εξαιρέσει που θα εκπνεύσουν ε, το 2018 και η δική σας αξιολόγηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν βρέθηκε λύση για τα non-cash collateral των συντεξοδοτικών ταμείων για τα οποία δόθηκαν αρχικά εξαιρέσει. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε για την αναθεώρηση τη σχετική νομοθεσία, πώ θα συνεργαστείτε με κεντρικού τραπεζίτε και εποπτικέ αρχέ για να βρεθεί μια λύση να διευκολύνει ε, την χρήση του Central Clearing από τα Ευρωπαϊκά Συνταξιδοτικά Ταμεία και τι κάλυψη προβλέπετε πέραν ε, του θέματο των συνταξιδοτικών ταμείων. Τώρα, για το θέμα του ΕΜΙΡ, της αναθεώρησης του κανονισμού αυτού, Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες από πέρυσι και είχαμε, ε, συγκεντρώσαμε πολλές παρατηρήσεις και ε, συστάσεις από πολλούς ενδιαφερομένους και είχαμε εκτεταμένες διαβουλεύσεις που εμπλούτησαν ε, τις γνώσεις μας. Πάντως, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο κανονισμός ΕΜΗΡ για τις υποδομές ευρωπαϊκών αγορών λειτουργεί καλά. Βέβαια κάποια θέματα όπως τα margin και τα καθαρά παράγωγα θα πρέπει να εφαρμοστούν. Πάντως η ουσία του κανονισμού είναι καλή. Θα επικεντρωθούμε ε, λοιπόν περισσότερο σε στοχευμένες προτάσεις που θα αφορούν θέματα υπερβάλλοντος ε, κανονιστικού άχθους ή την ανάγκη της αναλογικότητας. Στόχος μας είναι να προτείνουμε κάποιες τροπολογίες για τον κανονισμό ΕΜΙΡ στις αρχές του επόμενου έτους, προκειμένου να οριστικοποιήσουμε τους κανόνες πριν οι εξαιρέσεις για τις συντάξεις εκπνεύσουν στα μέσα του 2018. Συνεχίζονται επίσης ε, οι εργασίες για τις ε, υπόλοιπες αλλαγές. Γι' αυτό και είναι προ η συζήτηση αυτή, δεν μπορώ να δώσω πιο λεπτομεριακά σχόλια. Πάντως γνωρίζουμε το θέμα των εξαιρέσεων ε, για τα συνταξιοδοτικά ταμεία και εν ανάγκη ίσως χρειαστεί να παρατείνουμε τις ισχύουσες εξαιρέσεις. Ο Ερίκε Καλβέ Σαμπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έρχεται για μια ακόμη φορά στην Επιτροπή μας. Θα κάνω τέσσερις ε, ερωτήσεις. Κατευθείαν στο ψαχνό, χωρίς πολλές περικοκλάδες επεξηγηματικές. Πρώτο, εδώ και πολύ καιρό μας καθησυχάζεται ότι το ευρώ είναι εκτός κινδύνου, υπάρχει ασφάλεια, σταθερότητα από χρηματοπιστωτική άποψη, αλλά αυτό δεν φαίνεται καθαρά στις αγορές. Υπάρχει μια μόνιμη ανησυχία, κάτι που είναι αρνητικό. Και μάλιστα πολύ συχνά αυτή η ανησυχία προέρχεται από μια ε, έλλειψη διαφάνειας και πυγμής. Έχω κατά νου δύο υποθέσεις. Την Deutsche Bank, για παράδειγμα, που αμφισβητεί τη σοβαρότητα των προσωμιώσεων ακραίων καταστάσεων. Και φαίνεται ότι εφαρμόζονται διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανάλογα με το γιατί τη τράπεζα μιλάμε. Και όπως είπε και ο Διολίκολ Καπ, ε, ε, δεν μπορούμε να, ε, ξεγελάμε, μπορούμε να ξεγελάμε έναν για πολύ καιρό, αλλά όχι όλο τον κόσμο συνέχεια. Οπότε κάποιες φήμες που ακούγονται ε, για, και ανησυχίες για τις Ιταλικές τράπεζες. Καλύτερα να φτιάξουμε τον, τράβο, τον τάβρο από τα κέρατα και να εφαρμόσουμε μια διαφάνεια. Επίσης, τι κάνετε, τι γνώμη έχετε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον αντίκτυπο του Brexit σε ό,τι αφορά τη δυναμική και τον απαραίτητο ρυθμό ε, που πρέπει να δοθεί στην ε, ολοκλήρωση της ε, Ένωσης Κεφαλαγορών, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύης Καταθέσεων και ούτω καθεξής. Γιατί δεν είναι σωστό μια χώρα που έχει ένα πόδι μέσα και ένα πόδι έξω να μας παραμποδίζει ή να επιβραδύνει τις διαδικασίες. Το έχετε υπόψη σε αυτό, έχετε επίγνωση και το λαμβάνετε υπόψη σε εργασίες σας. Τέλος, τελευταία ερώτηση. Τι μπορείτε να μας πείτε για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την φερεγγιότητα των επιχειρήσεων. Ξέρω ότι βρίσκεται σε βάση διαβούλευση σε αυτό το θέμα. Έχετε κάποια πρόθεση, κάποιο όραμα, κάποιο προσανατολισμό για το θέμα αυτό για την περίφημη δεύτερη ευκαιρία που θέλουμε να δώσουμε και που είναι πολύ σημαντική για πολλές μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω εν συντομία να τις απαντήσω όλες. Ως προς την πρώτη ερώτηση τα αποτελέσματα των προσωμιώσεων ακραίων καταστάσεων στο τραπεζικό σύστημα. Τα αποτελέσματα είναι σαφή, ότι γενικώ το τραπεζικό σύστημα ε, έχει και καλύτερη κεφαλαιοποίηση και είναι σε πολύ καλύτερη φόρμα από ό,τι πριν από καμιά διετία. Βέβαια, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες αδυναμίες και φροντίζουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Αναφέρθηκατε σε συγκεκριμένες τράπεζες. Δεν πρόκειται να σχολιάσω την κατάσταση συγκεκριμένων τραπεζών. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μεθοδολογία των προσωμιώσεων κρέων καταστάσεων, τα stress test αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, οπότε καλύτερα να τα πείτε με την ΕΑΤ ποιε είναι οι μεθοδολογίε αυτών των προσωμιώσεων ακραίων καταστάσεων. Πάντω, γενικώ φαίνεται ότι οι τράπεζε πρέπει να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό του μοντέλο προκειμένου να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές και κανονιστικές αλλαγές και εξέλιξεις. Αναφέρεται και την κατάσταση του Ιταλικού τραπεζικού κλάδου. Έγινε κάποια πρόοδος τα τελευταία χρόνια προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των Ιταλικών τραπεζών και υπάρχει κάποια πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί μια τυπλοποίηση ενός τμήματο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και γίνονται διαβουλεύσεις και με τις Ιταλικές τράπεζες ενώ συνεργαζόμαστε στενά και με τις Ιταλικές αρχές για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Για τον αντίκτυπο του Brexit. Φυσικά είναι σημαντικό να είναι όλα τα κράτη-μέλη επικοδομητικά στην προσέγγιση της ε, για τους κανονισμούς του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Αλλά αυτό είναι ευρύτερο ζήτημα. Δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο κλάδο. Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο για την αφαιρεγγιότητα και τι θα προτείνουμε. Όσον θα προτείνουμε μια οδηγία ελάχιστης εναρμόνισης για την αναδιάρθρωση του βιώσιμου χρέους των επιχειρήσεων. Αυτό που είπατε δηλαδή, να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στις εταιρείες, στις επιχειρήσεις. Θα κατατεθεί ο ονόπο η σχετική πρόταση, αλλά θα αναλάβουμε και μια ευρύτερη πρωτοβουλία, τη συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών πλαισίων αφαιρεγκαιότητας που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη, ε, αναζητώντας τις καλύτερες ε, και πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις και εντοπίζοντας τα σημεία που χρειάζονται ε, μεταρρυθμίσεις. Θα ζητήσουμε πιο ακριβείς πληροφορίες από τα κράτη-μέλη για τα αποτελέσματα, δηλαδή τι χρέος έχει ανακτηθεί, πόσο γρήγορα διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες αφαιρεγκαιότητα και ούτω, ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντομπρόφσκης, ε, σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στην ε, Επιτροπή μας. Αναφερθήκατε στις προβλέψεις για την ανάπτυξη το 2017. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω ειδικότερα για τη χώρα μου την Ελλάδα. Έχω υπόψη μου μια δήλωσή σας πριν δύο μέρες ε, στο Eurogroup μιλήσατε για επιτυχία στην επίτευξη των φετινών δημοσιονομικών στόχων από την Ελλάδα σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα και κάνατε και κάποιες εκτιμήσεις εκ μέρους της Κομισιόν για το ύψος της ανάπτυξης της οικονομίας της Ελλάδας καθώς και για το πρωτογενές πλεόνασμα που υπάρχει ως στόχος το 2017. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις σας για το 2017 και για την πραγματική οικονομία και για τον, τα δημόσια οικονομικά. Και η δεύτερη μου ερώτηση, θα είμαι πολύ σύντομος, ο συνάδελφός σας, ο Επίτροπος Μοσκοβισή, επίσης προχθές επανέλαβε ότι θεωρεί αναγκαία και εφικτή μια ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, καθώς και μια συμφωνία για το χρέος, όπως έχει Περιγραφή τον Μάιο του 2016 με τη συμμετοχή και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και με απόφαση για βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυσης του χρέους μέσα στο 2016. Σημερίζεστε αυτή την εκτίμηση και εργάζεται η Κομισιόν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Για την κατάσταση στην ελληνική οικονομία, η προσδοκία μας είναι ότι η ελληνική οικονομία ήδη τώρα ε, έχει επανέλθει στην ε, ανάπτυξη ε, ανατρίμηνο μιλώντας Βεβαίως στο σύνολο του έτους ε, αναμένουμε 0,3% ύφεση αλλά μια οικονομική αύξηση 2,7% ισχυρή ανάπτυξη το επόμενο έτος. Οπότε η ελληνική οικονομία επιστρέφει στην ανάπτυξη. Και επίσης για τα δημοσιονομικά γνωρίζουμε ότι οι στόχοι του προγράμματος ε, έχουν τεθεί με έναν τρόπο διαρθρωμένο αλλά αναμένουμε ότι ήδη φέτος το έλλειμμα του προπολογισμού θα είναι κάτω από το 3%, θα είναι 2,5% του ΑΕΠ και θα συνεχίσει να μειώνεται στο 7% ίσως του χρόνου. Στο 1% με συγχωρείτε. Και όσον αφορά τον στόχο του, του διαρθρωτικού ισοζυγίου είναι 1,25% το ΕΠ και θεωρούμε ότι είναι απολύτως επιτεύξιμος. Κατόπιν, για τα μέτρα για το χρέος. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχαμε αναφέρει ήδη στο Eurogroup του Μαΐου. Τα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα και με βάση αυτό συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Οι συζητήσεις αυτές για το χρέος θα είναι μέρος των συζητήσεών μας στο πλαίσιο της δεύτερης ε, αυτής ε, αξιολόγησης. Βεβαίως ε, δεν είμαστε εμείς οι πιστωτές της Ελλάδας, όπου είναι οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης, οπότε αυτές τελικά θα αποφασίσουν, αλλά οπωσδήποτε η Κομισιόν θα παίξει τον ρόλο της για να διευκολύνει μια συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Σκοτ Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά να συγχαρώ τον Επιτροπό για όλα τα θέματα που ανέφερε το ευρύ, το φάσμα. Ήθελα να αναφερθώ στο Brexit. Θεωρούμε λοιπόν ένα δεδομένο ότι το Brexit θα χάσει την ιδιότητα του κράτους μέλους και θα αποτελεί πλέον τρίτη χώρα όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συνεπώς δεν θα μπορεί πλέον να επωφελείται από τις προβλέψεις για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της Ευρώπης, παρότι δεν ε, έχει προταθεί ε, δημοκρατική εποπτεία αυτή τη στιγμή που να καλύπτει συζητήσει. Ακούμε φήμε ότι κινούμαστε προ ένα σκληρό Brexit, το οποίο φυσικά εμένα με λυπεί ιδιαίτερο. Κάτι που σημαίνει ότι, αν μη τι άλλο, προτείνεται όχι μόνο να αναχωρήσουμε και από την ΕΟΧ, αλλά και την Τελωνιακή Ένωση. Πρόσφατα στο Bloomberg ο Μαρκ ανέφερε ότι σε περίπτωση hard Brexit ή soft Brexit όλα θα είναι δύσκολα και ο Γκαρνιά, ο ε, ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα μιας νέας ε, σχέσης πρότεινε μια διευθέτηση σχεδιασμένη ειδικά για αυτές. Οπότε η ερώτησή μου προς εσάς κύριε Επίτροπε είναι τι πιστεύετε ότι έχει στο νου του ω συμφωνία, κατά την άποψή σα, ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για την Ευρωπαϊκή Ενία Αγορά, αν κάνει μια τέτοια συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ήθελα να μάθω αν οι υπηρεσίε σα έχουν αναλάβει, έχουν ξεκινήσει ε, συζητήσει για οποιοδήποτε τέτοιο μέλλον, ε, ε, για οποιαδήποτε τέτοια μελλοντική συμφωνία. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι έχει επισημανθεί πολλές φορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από άλλους ε, ευρωπαίους ε, θεσμούς ότι οι τέσσερις ελευθερίες είναι ένα ενιαίο κομμάτι. Δεν μπορούμε να τις διαχωρίσουμε. Δεν μπορεί να διαλέγει ο καθένας ό,τι θέλει από τις τέσσερις ελευθερίες που αποτελούν το θεμέλιο της εσωτερικής μας αγοράς. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση. την οποία ακολουθούμε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δεσμευτούμε για πιο λεπτομερείς συζητήσεις, διότι και για αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε σαφής θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις μόνο αφού ενεργοποιηθεί το άρθρο 50. Δεν θα υπάρχουν διαπραγματεύσεις ή οτιδήποτε άλλο σχετικό πριν από αυτό. Οπότε τώρα το μπαλάκι είναι στο δικό σας γήπεδο όσον αφορά το άρθρο 50 και την ενεργοποίηση του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω τον Μάρκο Τζάνι, ο κύριος αννεμόντς. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η ομάδα μας δεν βλέπει γιατί πρέπει να είναι ε, συνδεδεμένες οι τέσσερις ε, Ούτως ή άλλως η Μεγάλη Βρετανία δεν ανήκε στην ε, ζώνη Σέγγεν. Λοιπόν, ελπίζω να κοιμηθήκατε καλά χτες το βράδυ, να ξεκουραστήκατε και να παρακολουθήσατε το πρωί την νέα κατάσταση. Και θα ε, σας ρωτάω γιατί Ξέρουμε όλοι πως ε, στην διεθνή οικονομία το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών μας οδηγεί μακριά από την τυποποίηση και το level playing field ως επιχείρημα για περισσότερη τυποποίηση στο σύστημα μέσω ακριβώς αυτής της διαδικασίας. Λοιπόν, Σα έλεγα εγώ θεωρούσα στα ζητήματα Βασιλείας 3 πως η διεθνοποίηση των διατάξεων για το κεφάλαιο, ανεξαρτήτως της συζήτηση ε, για την Ομοσπονδιακή Ευρώπη, την περαιτέρω ενοποίηση κτλ, πως η παγκοσμιοποίηση των διατάξεων για το κεφάλαιο ήταν ε, Αντίστοιχα με αυτούς οι οποίοι ε, ε, ήθελαν να πάνε ε, προς την μεριά των Αμερικανών, αλλά ακούγοντάς σας μάλλον έχω κάνει λάθος. Εσείς θέλετε μάλλον να πατήσουμε τον και να πάμε λιγορότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχω δίκαιο. Okay. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της Βασιλείας 3. Έχουμε αποκρισταλώσει τη γνώμη μας εδώ και πολύ καιρό και επιβεβαιώθηκε μάλιστα και δύο φορές από τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΕΚΟΦΗΝ του Ιουλίου αλλά και σε προηγούμενο ΕΚΟΦΗΝ. Όχι το τελευταίο, αλλά τα προηγούμενα. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να εμείνουμε στη Συμφωνία της Βασιλείας και η ολοκλήρωση της Βασιλείας 30 πρέπει να οδηγήσει σε σημαντική ε, συνολική αύξηση των κεφαλαϊκών απαιτήσεων. Επίσης, θα πρέπει να κρατήσουμε την ε, ευαισθησία του, του συστήματος ως προς τον κίνδυνο, ώστε οι τράπεζες να έχουν κίνητρα να επιλέγουν Λιγότερα ρηψοκίνδυνα επιχειρηματικά μοντέλα. Και αυτό ε, φαίνεται αντίστοιχα στις κεφαλαϊκές απαιτήσεις. Η προσέγγιση αυτή έτυχε ομόφωνης ε, υποδοχής στο Συμβούλιο Εκοφήν. και συζητήθηκε και στη Βασιλεία 3. Και μάλιστα ευελπιστούμε ότι θα, θα υλοποιηθεί και η συμφωνία προς τη διεκπαιρέωση της βασιλεστρία. Αύριο θα ψηφίσουμε και το σχετικό ψήφισμα για το σημείο αυτό, που κατά πάσα πιθανότητα θα ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τι αρχέ αυτέ. Μου έμεινε ένα λεπτό. Θα ήθελα να σας ε, πω να παρακολουθείτε τα όσα συμβαίνουν στην άλλη του, του Ατλαντικού. Μπορεί να μην αλλάξει επισήμω ακόμα η Βασιλεία αλλά μάλλον έχει αλλάξει ολόκληρη η ατμόσφαιρα όσον αφορά την διεθνή ολοκλήρωση σε αυτά τα πράγματα. Δεν να σχολιάσετε άλλο, όχι. Ωραία, ευχαριστούμε. Ο κύριος Οκμάρκ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε για την παρουσίαση σας εδώ σήμερα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε την ανάπτυξη. Διότι όπως είπατε, οι ευρωπαϊκές οικονομίες ε, παρουσιάζουν κάποιες πρόπτικες ανάπτυξης για του χρόνου, αλλά αυτή, είπατε, θα ε, βασίζεται σε μια ε, εξαιρετική νομισματική πολιτική, αρνητικά επιτόκια, κάποιοι θα έλεγαν υπερβολικά εξαιρετική διάφορα ε, νομισματικά μέτρα. Πόσο βιώσιμο πιστεύετε είναι όλο αυτό, γιατί υπάρχει και μια άλλη πλευρά του νομίσματος αυτού, ότι η νομισματική πολιτική θέτει σε κίνδυνο την κατάσταση, διότι μπορεί να δημιουργήσει χρηματοπιστήτικη φούσκα. Η ανάπτυξη λοιπόν που παρατηρούμε πόσο κομμάτι αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση τη ανταγωνιστικότητα βάσει μεταρρυθμίσεων και πόσο κομμάτι αυτή αντιστοιχεί σε μια νομισματική πολιτική που μακροπρόθεσμα δεν είναι βιώσιμη. Το λέω αυτό διότι πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να γίνει μια αξιολόγηση αυτού ώστε να μπορούμε να κρίνουμε ποια θα είναι η μεταρρυθμιστική πολιτική στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό όμως επίσης και για να έχουμε μια γενικότερη εικόνα του πόσο εύθραυστες είναι οι οικονομίες μας δεδομένου του νέου Αμερικανού Προέδρου όπως μπορεί να δημιουργήσει διάφορους φραγμούς για τις ε, διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Πόσο βιώσιμη λοιπόν είναι η ανάπτυξη. Πώς βλέπετε τους κινδύνους της νομισματικής πολιτικής και σε ποιο βαθμό πιστεύετε έχουμε κάνει μεταρρυθμίσεις όπως θα έπρεπε Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ερωτήσεις. Λοιπόν, για το πόσο βιώσιμη είναι η, οικονομική μας ανάκαμψη, είναι κάτι που τονίζει η Κομισιόν, ότι η οικονομική ανάπτυξη έχουμε φέτος, αλλά μέτριο επίπεδο. Χρειάζεται να την ενισχύσουμε και να την καταστήσουμε πιο βιώσιμη. Όσον αφορά την νομισματική πολιτική, κάτι που τόνισε ε, ο ίδιος ο Μαριο Ντράγκη, είναι αδύνατο να επιλύσουμε διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας με την νομισματική πολιτική μόνο. Η νομισματική πολιτική βοηθά να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίσουν χρόνο τα κράτη-μέλη, αλλά ο χρόνος αυτός θα πρέπει να αξιοποιηθεί σοφά ώστε να υλοποιηθούν πραγματικά οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό το λόγο συζητάμε τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε ορίσει τρεις προτεραιότητες. Ενίσχυση των επενδύσεων, διότι είναι σαφώ ότι έχουμε έλλειμμα επενδύσεων, ε, το οποίο είναι βραχυπρόθεσμο πρόβλημα που θα επηρεάσει και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές αρνητικά. Χρειαζόμαστε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να εξυγχρονίσουμε τις οικονομίες μας και χρειαζόμαστε και δημοσιονομικά υπεύθυνε πολιτικές, διότι δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς, ε, μη βιω... βιώσιμα δημοσιοοικονομικά. Αυτά τα τρία στοιχεία λοιπόν είναι εξίσου σημαντικά. Το ίδιο και τα στοιχεία της επισκόπηση επισκόπησης της ανάπτυξης που εξακολουθούν να ισχύουν ε, και για την προετοιμασία της επόμενης ε, ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης. Πώς προχωρά λοιπόν αυτό το θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων. Προχωρά θα έλεγα, αλλά φυσικά πάντα ευχόμαστε καλύτερη πρόοδο. Για παράδειγμα, όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων κατά χώρα, ε, σύμφωνα με τις δικές μας αξιολογήσεις, έχουμε περιορισμένη ή κάποια πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων αυτών κατά χώρα που έχουμε εκδώσει. Αυτό δείχνει σαφώς ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα σε θέματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Είναι κάτι που εμείς επισημαίνουμε έντονα και στις συζητήσεις μας με τα κράτη-μέλη το ότι η εφαρμογή των συστάσεων κατά χώρα πρέπει να βελτιωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νίνα Γκίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίσατε κύριε Αντιπρόεδρε, τον Οκτώβριο. Κάνετε μια ομιλία στην ΙΟΚΙ και είπατε, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις ε, χωρίς ε, άροντα τα διασυνοριακά εμπόδια. Καταπληκτικά αλλά γίνει η κοινή νομισματική ένωση, ε, η ένωση του φελεγόρων στην οικονομία. Πραγματικότητα χρειάζεστε τη συνεργασία του τομέα, ε, του χρηματοπιστωτικού τομέα και μεγάλο κομμάτι που βρίσκεται στο Λονδίνο και κάποιοι λένε ότι η Κομισιόν έχει χάσει το όρομα, δεν ξέρει σαφώς πώς πρέπει να κινηθεί. Και αντίθετα εστιάζεται σε τεχνικά προβλήματα όπως το καθεστώς ε, ε ισοδυναμίας να σας ρωτήσω πώς θα τα προχωρήσουμε όταν θα πρέπει να εστιαζόμαστε στο στόχο της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας και να χρησιμοποιούμε ό,τι μπορούμε ως επιλογές για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Φαίνεται να κινούμαστε προς την αντίθετη κατεύθυνση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εικόνα ότι εφαρμόζει προστατευτισμό η Ευρώπη. και είναι σαν να επιτρέπουμε τα αποτελέσματα του Βρετανικού Δημοψηφίσματος να μας εκτροχιάζουν από τον αρχικό στόχο. Ξέρετε, φαίνεται σαν να παρεκκλίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις υποσχέσεις του Γιούνκερ πριν από 2,5 χρόνια και απομένουν μόλις 2,5 χρόνια για την Επιτροπή αυτή. Τώρα, δεδομένων αυτών των χρονικών προθεσμιών, δεν γνωρίζουμε ακριβώ πώ θα κινηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο τελικά και που θα βρίσκεται. Οπότε θεωρώ ότι είναι επίγον η Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρει αποτελέσματα, δεδομένου ότι υπάρχουν εκλογέ στη Γερμανία, στη Γαλλία. Και μόλις εξελέγει και ο πιο προστατευτικός πρόεδρος της ΗΠΑ, βρισκόμαστε σε επικίνδυνα νερά. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να επιτύχουμε την επιτεύξη των αποτελεσμάτων και των στόχων. Δεύτερον, ε, συμμερίζομαι τα σχόλιά σας για τον τραπεζικό τομέα και εγώ ανησυχώ για τι πιθανέ αρνητικέ επιπτώσει των συζητήσεων για το Βασιλεία ε, στην οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανώ τι αρνητικέ επιπτώσει για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και τη χρηματοδότηση των υποδομών. Και ανησυχώ ιδιαίτερα για την ταχεία ανάληψη ε, λήψη αποφάσεων και την έλλειψη διαφάνεια στην όλη διαδικασία. Ανησυχείτε και εσεί το ίδιο. Τι εγγύησει μπορείτε να δώσετε ότι οι προτάσει που θα παρουσιάσετε σε εμά μετά βάσει των συστάσεων της Βασιλείας θα είναι αναλογικές και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τους κοινού μας στόχους για δημιουργία ανάπτυξη και θέσεων εργασία. Ευχαριστώ. Ε, Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Καταρχήν για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Ήταν μια από τις πρώτες αντιδράσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το δημοψήφισμα για το Brexit. Συντάξαμε ανακοίνωση για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, προσπαθώντας να επιταχύνουμε το έργο όπου μπορούσαμε. Και μάλιστα ακριβώς αποσαφηνήσαμε το γεγονός ότι η προοπτική αυτή της μεγαλύτερης ε, κεφαλαγοράς να, να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά την ανάγκη της Ένωσης Κεφαλαγορών ακόμη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή την προσέγγιση θα ακολουθήσουμε και στο μέλλον. Θα δούμε πώς θα υλοποιήσουμε ε, τους στόχους μας. Καταρχήν θα πρέπει να καταλήξουμε ε, σε συμφωνία στο, στην πρώτη δέσμη προτάσεων που έχουμε ήδη καταθέσει και εξετάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί πολύ, πολλά νομοθετικά θέματα έχουν ήδη διεκπαιρεωθεί στο Συμβούλιο, έχει καταλήξει συμφωνία εδώ και ένα χρόνο. Περιμένουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τώρα για να ξεκινήσουμε τους τριμερείς διαλόγους. Και σίγουρα μπορούμε σε ορισμένους τομείς να επικεντρωθούμε για να επισπεύσουμε τις εργασίες. Κάτι άλλο που θα εξετάσουμε σε ό,τι αφορά την πρόταση CRR είναι ο αντίκτυπός του στα μακροπρόθεσμα θέματα των οικονομικών, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις υποδομέ. Οπότε ε, οι δεσμεύσεις μας ε, δεν έχουν ε, υποβαθμιστεί. Το αντίθετο, είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι από ποτέ να ολοκληρώσουμε την Ένωση Αγορών. Σε ό,τι αφορά τώρα τις τράπεζες και τα αποτελέσματα της Βασιλείας, επαναλαμβάνω, η θέση στην οποία καταλήξαμε φαίνεται ότι είναι κοινή αποδοχή. Στόχος μας είναι μια καλή συμφωνία στη Βασιλεία και σίγουρα αν έχουμε νέα φωνή, θα έχουμε και ισχυρότερη θέση. Θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να επιδείξουμε ενότητα. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απλώς παρατηρητή στη Βασιλεία, όχι μέλος. Αλλά προσπαθούμε να συντονίσουμε τη θέση των κρατών μελών, ώστε να εκφράζουμε μια νέα θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονισμένη στις διαπραγματεύσεις, μια συμπαγή θέση είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε καλή συμφωνία στη Βασιλεία. Μια καλή συμφωνία που θα μπορέσουμε στη συνέχεια να εφαρμόσουμε. Στην πρόταση, στις ανακοινώσεις μας, λαμβάνουμε υπόψη τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες και μεταξύ άλλων και την ανάγκη της χρηματοδότησης της ευρύτερης οικονομίας και αυτό αποτελεί σημαντικό κριτήριο κατά την, το σχεδιασμό των αποφάσεων. Πρώτα όμως χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη συμφωνία στη Βασιλεία. Σας ευχαριστώ, Χωσέ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλωσορίζω και εγώ τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα υποβάλω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταρχήν, πώς αξιολογείτε την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Δεύτερον, πώς βλέπετε την ανάπτυξη στην πατρίδα μου, την Πορτογαλία. Τρίτον, πώς αξιολογείτε τον προϋπολογισμό του 2017 και πώς εξηγείτε τις ε, σημαντικές διαφορές που υπάρχουν στις προσωμιώσεις, ε, τις εκτιμήσεις ε, και τους υπολογισμούς μεταξύ της πρώτας προϋπολογισμού και της αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης ποιες είναι οι συστάσεις σας ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί σε ρυθμούς ανάπτυξης και η Πορτογαλία το ίδιο και ποιες είναι οι συγκεκριμένες συστάσεις για την Πορτογαλία και για τον προϋπολογισμό του 2017. Ευχαριστώ. Πρώτα, για την ανάπτυξη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προβλέψεις ανάπτυξης για την Ευρωζώνη. Όπως σας είπα είναι μετριοπαθής η οικονομική ανάκαμψη, αλλά συνεχίζεται. Και γι' αυτό αναβαθμίσαμε ελαφρώς τις εκτιμήσεις μας ε, για την ανάπτυξη φέτος. Αλλά τις μειώσαμε κάπως για του χρόνου. Ήταν πάντως σχετικά μικρές οι αλλαγές, 0,1-0,2%. Οπότε η γενικότερη εικόνα παραμένει αμετάβλητη συνεχίζουμε να έχουμε μια ναι μέτρια αλλά εμφανή ανάπτυξη και ελπίζουμε να συνεχιστεί και προσπαθούμε να το επιδιώξουμε. Τώρα, η οικονομική ανάπτυξη της Πορτογαλίας ε, θα είναι κάτω από το κοινοτικό μεσοόρο, 0,1% για φέτος και 1,2% για το χρόνο. Τώρα, ποιες ε, είναι οι συστάσεις μας για την Πορτογαλία και στα δημοσιονομικά. Θα σας συμβουλεύαμε καταρχήν να κρατήσετε σταθερή την πορεία σας, να μην ακυρώσετε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν και σε αυτό το πλαίσιο της αυξανόμενης αβεβαιότητας που επικρατεί είναι ιδιαίτερο σημαντικό να παραμείνουμε προνοητικοί, επιφυλακτικοί στις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές μας. Γιατί όταν υπάρχει μια γενική αβεβαιότητα, υπάρχει ένα φυσικό φαινόμενο της αναζήτησης ε, της ασφάλειας, κάτι που ε, αφήνει εκτεθειμένες τις περιφερειακές οικονομίες. Γι' αυτό σε αυτό το πλαίσιο είναι σωστό είναι σημαντικό να στείλουμε τα σωστά μηνύματα. Για παράδειγμα για την Πορτογαλία ότι κρατά τη δημοσιονομική της τροχιά και μένει στις δημοσιονομικές ε, μεταρρυθμίσεις της. Ο κύριος Φερνάντες, ο άλλος Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο τον ε, για την παρουσία του εδώ. Ενώνω και εγώ τα συγχαρητήριά μου σε αυτά του Πάολο Σάλμπα ε, για την ε, ενίσχυση του χαρτοφυλακίου σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το ΕΔΙΣ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αγγίσης Καταθέσεων. Πριν από λίγες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το, τη μελέτη επιπτώσεων, τη μελέτη αντικτύπου του ΕΔΙΣ. Ε, ακούστηκε όμως εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ελάχιστες διαφορές βλέπει η μελέτη αντικτύπου μεταξύ ενός συστήματος ε, πλήρους ασφάλισης και συστήματος αντασφάλισης. Εγώ βλέπω αισθητέ διαφορές, αλλά θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση. Σήμερα το πρωί είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί της εκθέσεως ε, της Έστερ Ντελάνκε, που είναι η συγκίτρια για το θέμα αυτό. Οι ε, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, δυστυχώ δεν είχαν χρόνο να λάβουν μέρο στη συζήτηση, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η αρχική σας αξιολόγηση της έκθεσης Λάγκε, μια και το πρωί οι συνεργάτες σας δεν είχαν την ευκαιρία να λάβουν το λόγο στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ε, first... Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα για τη δομή των προτάσεων για το ένδυστο ε, σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Αρχικά η Κομισιόν είχε προτείνει να ξεκινήσουμε με μια προσέγγιση αντασφάλισης που σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα τα κράτη-μέλη θα χρησιμοποιήσουν τα εθνικά του συστήματα εγγυήσεων καταθέσεων πριν προσφύγουν στα ευρωπαϊκά και μετά πάμε στην συνασφάλιση που σημαίνει ότι κάποιο τμήμα των απολειών ε, θα ε, τα ποσά δηλαδή θα εκταμιεύονται αμέσως από ένα ευρωπαϊκό σύστημα και αυξάνεται το ποσοστό αυτό από το 20-30% και μετά πάμε στην πλήρη ασφάλιση. Βεβαίω είμαστε ακόμα ανοιχτοί στο να συζητήσουμε την ακριβή τροχιά, πώς θα φτάσουμε από την τρέχουσα κατάσταση στο, στην πλήρη ασφάλιση σύμφωνα με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Όσον αφορά τις αντιδράσεις Κομισιόν στο σχέδιο έκθεσης της Εστέρ Ντελάνγκε, όπως είπα μόλις δημοσιεύτηκε, οπότε αξιολογούμε ακόμα τις διάφορες λεπτομέρειες. και κοιτάμε μετά τι θα γίνει με την αρχική πρόταση της Κομισιόν και το πώς ταιριάζουν αυτά τα δύο. Αλλά όπως είπα και στην προηγούμενη ερώτηση, οπωσδήποτε εμείς ως Κομισιόν είμαστε στην ε, ε, διάθεσή σας για να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές λύσεις για να έχουμε μια συμφωνία για το σύστημα ασφάλισης καταθέσεων. Βεβαίω, σε κάθε περίπτωση η έκθεση αυτή ε, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα στην Επιτροπή. Ακριβώς, λέει ο πρόεδρο. Οπότε, πριν τον συμβασμό πρέπει να καταλήξει μια θέση στο Κοινοβούλιο. Το... Αυτό κάνουμε. Λοιπόν, και πάλι, Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες, ε, δεύτερη ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, φάνηκε από τη συντριπτική πλειοψήφια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θέλουμε αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πρώτο καθεδρία του κράτους δικαίου, αποφύγη των διακρίσεων και όπως λέει και το βιβλίο του Ολάντ, ένας πρόεδρος δεν θα πρέπει να λέει κάτι τέτοιο. Και σε αυτό το βιβλίο λέει ο Ολάντ ότι υπάρχει συμφωνία ώστε η Γαλλία να μην έχει την ανάγκη να σεβαστεί και να τηρήσει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ερωτώ λοιπόν, ε, κάποια δυσφορία ως προς την εφαρμογή αυτού του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, πως δεν υπήρχε ποτέ αυτή η συμφωνία γιατί θα ήταν παραβίαση της νομοθεσίας ε, ε να εφαρμόζεται επιλεκτικά από ορισμένε χώρες και αυτό πραγματικά θα ήταν η απευκταία διακριτική μεταχείριση που είπα. Uh, ναι. Ας είμαστε σαφείς. Όλες οι χώρες πρέπει να σέβονται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και αυτό ισχύει εξίσου και για τη Γαλλία. Οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω για, για κάποιες συγκεκριμένες αναφορές που έγιναν σε βιβλία. Αυτή είναι η θέση της Κομισιόν, είναι σαφής και όσον αφορά συγκεκριμένα την συμμόρφωση της Γαλλίας με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είχαμε πολύ έντονο διάλογο με την κυβέρνηση από την αρχή της θητείας αυτής της Επιτροπής και το τονίζουμε ξανά και ξανά ότι η Γαλλία πρέπει να διορθώσει το υπερβολικό έλλειμμα σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, δηλαδή το επόμενο έτος. έχουμε την δέσμευση της γαλλικής κυβέρνησης ότι πράγματι θα επιμείνουν και βλέπουμε ότι το σχέδιο προϋπολογισμού ακριβώς καταρτίζεται με στόχο να διορθωθεί το υπερβολικό έλλειμμα. Αν βεβαίω θα χρειαστεί να συζητήσουμε τον αντίκτυπο συγκεκριμένων μέτρων, στο σχέδιο προπολογισμού της Γαλλίας, αλλά υπάρχει η δέσμευση της κυβέρνησης και ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθούμε προσεκτικά το να σεβαστεί η κυβέρνηση αυτή τη δέσμευσή της. Ευχαριστώ. Πέντρο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλώς ήρθατε. Δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη έχει να κάνει με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στους ισολογισμούς των τραπεζών. Βεβαίως το συζητάμε εδώ και καιρό αυτό το θέμα. Στις ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης πέρσι τον Νοέμβριο η Κομισιόν είπε ότι ε, θεωρεί, ε, εξετάζει με συγχωρείτε, μια πρόταση που θα αντιμετωπίσει ακριβώς το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό το οποίο μας είπατε είναι ότι ασκείται πίεση σε αρκετά κρατημέλη μέσω των συστάσεων αναχώρα και ότι αναζητείται συγκεκριμένες ε, λύσεις προσαρμοσμένες στην κάθε χώρα, ειδικά με τις Ιταλικές αρχές. Θα ε, ήθελα να μας πείτε κάποια συγκεκριμένα πράγματα για την πρόταση που θα υποβάλει η Κομισιόν, εάν υποβάλει, και αν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι τέτοιες προτάσεις περιλαμβάνουν τα οχήματα ειδικού σκοπού, όπως λέγονται, που δημιουργούν τα κράτη-μέλη για να απορροφήσουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να φύγουν αυτά από τους ισολογισμούς των τραπεζών. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με την αξιοπιστία του συστήματος Bailin στην ατζέντα της ε, Κομισιόν για την Τραπεζική Ένωση, πέρα από το ζήτημα των Μπέιλιν και των λεγόμενων ελάχιστων απαιτήσεων για τις, ε, για τις αποδεκτές υποχρεώσεις. Υπήρχε η πρόταση για την συνολική δυνατότητα απορρόφησης ζημιών να εφαρμοστεί δηλαδή πλήρως ε, η διεθνής προδιαγραφή. Θα ήθελα να γνωρίζω αν επιβεβαιώνεται αυτό το χρονοδιάγραμμα και αν ισχύει αυτό ποιο μοντέλο εξετάζει η Κομισιόν. Συγκεκριμένα σκέφτεστε να προτείνετε κάποια συγχώνευση μεταξύ του MREL και του TILAC. Για την πρώτη ερώτηση, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όντως οι συνθήκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα και το νομοθετικό πλαίσιο επίσης. Παρόλα αυτά, εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και τις Εθνικές Εποπτικές ε, αρχές για το πώς θα μπορέσουν οι χώρες να αντιμετωπίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά βεβαίως είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Και βλέπουμε ότι πολλά κράτη-μέλη το αντιμετωπίζουν με διάφορους ε, τρόπους. Ε, πολλά κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα ανοίγουν τις αγορές μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά ε, φτιάχνουν τις λεγόμενες bad banks αλλά όπως η τράπεζα αλλάζουν τους κανόνες για το ποιος θα υπομίζεται τα βάρη ή άλλα πουλάνε τα μη εξυπηρετούμενα βάρη σε τιμές αγοράς όπως η Ουγγαρία. Εξετάζουμε λοιπόν την ε, εμπειρία του Ιταλικού συστήματος τιτλοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και και κοιτάμε και τις ε, συστάσεις ε, αναχώρα για να βρούμε λύσεις προσαρμοσμένες στην κάθε χώρα. Οπότε συνεχίζεται αυτή η δουλειά και συνεργαζόμαστε με τα κρατημέλη στην ε, Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών για να έχουμε μια συνολική ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και όλες αυτές τις ε, πτυχές. Ε, είναι λοιπόν μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Επίσης, ναι, πράγματι θα κατεβάσουμε μια πρόταση για το TILAC και στους επόμενους μήνες θα ανταποκριθούμε στις ε, διεθνείς μας ε, δεσμεύσεις. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο καθεστώτων, καθώς το ΤΙΛΑΚ ε, συμφωνεί με την Διεθνή Συμφωνία για τις παγκόσμια σημαντικές συστημικές τράπεζες, ενώ το ΕΜΡΕΛ ισχύει για όλες τις τράπεζες, αλλά εν θα πρέπει να φροντίσουμε αυτά να συνδυάζονται και να μην υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των δύο πλαισίων. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο ακόμα το επεξεργαζόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Πιτρόπε. Θα ήθελα να μιλήσουμε για το αρχείο Μηφικ 2 το οποίο ψηφίστηκε βέβαια αρχικά το 2014 και μετά από αίτημα της Κομισιόν εδώ η Επιτροπή ενέκρινε ε, προθεσμία ε, υλοποίησης για ένα έτος πέρυσι λόγω καθυστερήσεων θα συζητούσαμε τα δύο κρεμόντα ε, αριθμιστικά πρότυπα για διάφορε εξαιρέσει και η πλειοψηφία σε εκείνη τη συνάντηση κάλεσε για ε, γρήγορη, για γρήγορη υιοθέτηση ώστε να γίνει υλοποίηση τον Ιανουάριο του 2018. Έχετε κάποια ιδέα, θα είναι δυνατόν να υιοθετηθούν αυτά τα RTS πριν τα τέλη του έτου ή προβλέπετε να ξαναέρθετε εδώ και να μα ξαναζητήσετε παράτηση τη προθεσμία για το ε, κείμενο του ΠΕΔΟΕΝΑ, 1. Όπως γνωρίζετε, στην περίπτωση του MIFID 2 είχαμε ήδη καθυστέρηση, οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε περαιτέρω καθυστερήσεις. Πιστεύουμε ότι είναι απόλυτος εφικτό. Ελπίζουμε λοιπόν να υιοθετηθούν τα δύο απομένοντα RTS για τα commodity derivatives σύντομα εφόσον υπάρχει ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για το ΜΕΦΙΤ που αρχίζει να, να ξεκινήσει το ΜΕΦΙΤ ε, στις αρχές του 2018. Το RTS ε, για τα όρια θέσεων είναι πιθανώς αυτό που προσέλξε περισσότερες συζητήσεις. Όπως συζητήσαμε σε μια συνάντηση που αφιερώθηκε σε αυτό το ζήτημα η εκτίμηση της Επιτροπής ήταν ότι η πρόταση του ε, είναι ισορροπημένη αλλά ε, ακούσαμε και τις απόψεις του Κοινοβουλίου οπότε εξετάσουμε τον καλύτερο τρόπο θα, με τον οποίο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε για τις μέγιστες εκθέσεις για τα όρια έκθεσης ε, για προϊόντα διατροφής αλλά είναι σημαντικό να επιτύχουμε και μία ε, ισορροπία εδώ, γιατί αφενός προσπαθούμε να ε, καταπολεμήσουμε την κερδοφορία, την ε, κερδοσκοπία, συγγνώμη, αλλά απ' την άλλη ακούμε από τους οργανισμούς των γεωργών ότι η πρότασή μας δημιουργεί προβλήματα σε αυτούς. Δεν τους δημιουργεί εμπόδια στις δραστηριότητες τους. ουσιαστικά στο να κάνουν τη δουλειά τους. Ε, παρεμποδίζει τις εργασίες τους όλο αυτό το σύστημα με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα πρώτων ελαιών Οπότε, ε, βασικών εμπορευμάτων, συγγνώμη, και δημιουργεί κινδύνου και για αυτού. Οπότε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ε, στι νέες αυτές προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση το μελετάμε αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε και εδώ μια καλή ισορροπία. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά θα επανέλθουμε και εδώ στο σημείο αυτό ως κοινοβούλιο. Θα σας στείλουμε τα σχόλια μας πολύ σύντομα. Είναι πολύ σημαντικό φυσικά να καταφέρουμε και να, να προβλέψουμε να προβλέψουμε να μην υπάρχουν υπερβολικά πολλέ ενστάσει. γι' αυτό είναι σαφέ ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε εμεί τη δική μα εκτίμηση, λαμβάνοντα υπόψη και την τελευταία πρόταση ε, για τη ρυθμίση των λεπτομεριών αυτού του στοιχείου που είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και πολύ περίπλοκο διότι υπάρχει κάποια ε, ε, εξαίρεση για το hedging ούτως ή άλλως οπότε πρέπει να δούμε πώς επηρεάζονται διάφορες κατηγορίες αγορών. Ερβάνς Μπερές, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, ήθελα να σας ρωτήσω ε, όσον αφορά τη συγχώνευση του Λονδρέζικου Χρηματιστηρίου. Αν χρησιμοποιώ το λάθος μικρόφωνο, λέει ο Μιλήτρια. Λοιπόν, κύριε Επίτροπε, κύριε Αντιπρόεδρε, να σας ρωτήσω για τη συγχώνευση του Λονδρέζικου Χρηματιστηρίου και της Deutsche Burs. Η συναδελφός σας, κυρία Φεστάγκερ, έχει κληθεί να εκφέρει απόψη για το θέματα ανταγωνισμού και έχει πει ότι θα αναλύσει αυτή την ε, δράση συγχώνευσης ανεξάρτητα από το Brexit. Λοιπόν, όσον αφορά αυτή τη συγχώνευση, τίθεται ένα θέμα διαγωνισμού πολύ σημαντικό, πολύ ευαίσθητο. Αλλά υπάρχουν και άλλε δύο πτυχέ στην υπόθεση αυτή που θα πρέπει να εξεταστούν ε, το ίδιο διεξοδικά. Ένα ρυθμιστικό ζήτημα και ένα ζήτημα εποπτεία. Και μετά υπάρχει το γενικότερο πλαίσιο με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί η κυρία Βεστάκερ ε, αλλά όπου έκανε σαν να μην υπάρχει, αλλά το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Λοιπόν, αν αυτή η συγχώνευση λάβει χώρα, θα είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση σε θέματα υποδομής θα αντιστοιχεί σε 25 δισεκατομμύρια χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε τέτοια κλίμακα σήμερα στην Ευρώπη. Θα βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου θα συζητάμε αφενός για το Brexit και θα λέμε πρέπει να τηρούνται οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς και θα έχουμε μια, την ύπαρξη μια τέτοια επιχείρηση, ε, τέτοιου κλίμακα ε, και τόσο συστημικού χαρακτήρα. Από άψη ρυθμιστική, η συμφωνία που συνάφθηκε και όπως έγινε δεκτή από το Λονδίνο βασίζεται στο γεγονός ότι η ρυθμιστική αρχή θα έχει έδρα στο Λονδίνο. Για να υπάρχει λοιπόν ισοδυναμία θα πρέπει να υπάρχει κάτι αντίστοιχο του ΕΜΗΡ ένας κανονισμός που τελικά παραπέμπει στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και από ό,τι κατάλαβα για το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό αποτελεί πραγματικά πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά το ζήτημα της εποπτείας ε, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε μια δημιουργία επιχείρησης απόλυτα συστημικής η οποία θα διαφεύγει από την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς ε, βλέπει η Κομισιόν το φάκελο αυτό ολόκληρο, όχι μόνο για θέματα ανταγωνισμού, θέμα το οποίο δεν είναι αρκετό για να αναλύσουμε πλήρως το διακύβευμα για τις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως προκύπτει από μια τέτοια συγχώνευση. Well, uh, uh... Όντως, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία συγχώνευσης ε, του Λονδρέζικου με το Γερμανικό Χρηματιστήριο, είναι ένα θέμα που για το οποίο έχει επιληφθεί η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και η Επίτροπος Βερστέγκερ. Ε, αξιολογείται η συγχώνευση ε, ακόμη. Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Και συμφωνώ απόλυτα ότι δεν υπάρχουν μόνο πτυχές ανταγωνισμού, αλλά και κίνδυνο συγκέντρωσης. Και αυτό κυρίως εξετάζει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Αλλά υπάρχουν και θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αλλά και κάποια ζητήματα ρυθμιστικά. Και σίγουρα και άλλη Γενική Διεύθυνση παρέχει πληροφορίες για τις υπόλοιπες πτυχές. Πάντως ε, η απόφαση θα ληφθεί σε τελική ανάλυση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Και επί του παρόντος δεν μπορώ να κάνω άλλα σχόλια, γιατί συνεχίζεται η εξέταση. Έχετε και συμπληρωματική ερώτηση ολοκληρώσατε. Ευχαριστώ για την απάντηση κύριε Αντιπρόεδρε, Πρόεδρε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν με ικανοποιεί η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Και γι' αυτό πιστεύω ότι εσείς ως αντιπρόεδρος, ίσως και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Γιούνκερ, θα πρέπει να εξετάσουν αυτά τα θέματα. Γιατί ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος. Και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κυρία Φερστάγκερ για να διερευνήσει τα ζητήματα ανταγωνισμού αλλά δεν έχει κανένα λόγο και δεν έχει καν αρμοδιότητα να εξετάσει η κυρία Βερστάγκερ τα ρυθμιστικά ζητήματα ή τον κίνδυνο στη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι εσείς ως αρμόδιος αντιπρόεδρος για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών θα μπορούσατε να ζητήσετε είτε την γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας ε, είτε τη γνώμη της ε, Επιτροπής, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου για τα θέματα αυτά. Ναι, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που υπερβαίνουν τα, τις αμυγείς πτυχές του ανταγωνισμού. Και αυτό εξετάζουμε επί του παρόντος για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Και σημειώνουμε φυσικά προσεκτικά τις ανησυχίες σας για να δούμε πώς θα διασκεδαστούν. Ο κύριος Τόιρερ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επίτροπος Βεστάγκερ μόλις αναφέρθηκε. Στο πλαίσιο αυτό είδαμε πως παραδείγματος χάρη μετά την απόφαση της ε, Κομισιόν ε, για την Ιρλανδία και την Apple ε, απευθύνθηκαν ε, στην Αμερικανική κυβέρνηση για να στραφεί κατά της Κομισιόν στο θέμα της Βασιλείας. Επίσης η Αμερικανική κυβέρνηση εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Αμερικανικής οικονομίας και από τις συζητήσεις έχει κανείς την εντύπωση πως η ΙΠΑ επιδεικνύουν ε, μια στάση απέναντι στις ευρωπαϊκές τράπεζες ε, που λένε ότι έχετε τόσο λίγο κεφάλαιο, τόσο λίγα κέρδη, από πού θα προκύψει ε, η κεφαλαιοποίηση και βέβαιως θεωρούν ότι αν μειωθούν σε μέγεθος τόσο ώστε να θεωρούνται υγιείς, θα υπάρξει και ένα μερίδιο της αγοράς που θα απελευθερωθεί και θα μπορέσουν έτσι να διεισδύσουν αμερικανικές εταιρείες και με βάση τα όσα ακούσαμε σήμερα από τις δηλώσεις Τραμπ America First και την ενίσχυση των ΗΠΑ, τίθεται το ζήτημα ξανά. Μήπως έχει φτάσει η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να, μια, κάνει μια αξιολόγηση για το εάν τα έχουμε, έχουμε προχωρήσει σε πολύ αυστηρή ρύθμιση στον τομέα των τραπεζών, πως πρέπει να αφήσουμε λίγο περιθώριο κερδοφορίας και να Έχουμε επίσης και μια διαφορετική επικοινωνιακή στρατηγική. Βλέπουμε με την Apple πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι μπορεί να φανεί ισχυρή και στιβαρή και τα κράτη-μέλη επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μιλάνε με μια φωνή και τότε είναι δύσκολο βεβαίως να υπάρξει ευρωπαϊκή θέση. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να ακολουθεί και μια άλλη επικοινωνιακή ε, στρατηγική. Σας ευχαριστώ. Ναι. Πολλές ερωτήσεις. Να φερθώ σύντομα στην περίπτωση της Apple γιατί πράγματι ήταν μία περίπτωση κρατικών ενισχύσεων και επιλεκτικής μεταχείρισης ε, μέσω των φορολογικών αποφάσεων και κατέληξε έτσι να πληρώνει πολύ ε, χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές από την συνήθις ε, εταιρική φορολογία στην Ισλανδία και ακριβώς αυτή η πτυχή της επιλεκτικότητας ήταν αυτή η ε, οποία ήταν ο πυρήνας αυτής της απόφασης και βλέπουμε ότι συχνά παρουσιάζεται ως μία απόφαση φορολογικής πολιτικής ότι είμαστε κατά των φορολογικών συντελεστών της Ιρλανδίας. Όχι. Αντιθέτως, η Κομισιόν λέει ότι η Apple θα πρέπει να πληρώσει ε, τον κανονικό φορολογικό συντελεστή για τις εταιρείες στην Ιρλανδία. Και για τη Βασιλεία Ήδη έχω σχολιάσει δύο φορές, δεν έχω πολλά να προσθέσω. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε με μία φωνή στην Βασιλεία. Και προς ε, αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε τώρα για το θέμα του εάν έχουμε κάποια υπερβολική ρύθμιση. Αυτός ακριβώς ε, ήταν ο στόχος μας όταν ζητήσαμε στοιχεία, ακριβώς να εξετάσουμε αυτές τις ε, πτυχές για να δούμε τι σορευτικό αποτέλεσμα έχουν όλα τα μέτρα τα οποία εγκρίθηκαν ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης, να αξιολογήσουμε δηλαδή πως τα ίδια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με λιγότερο επιβαρυντικά μέτρα και πιο αναλογικά, ειδικά όταν μιλάμε για μικρότερες ε, εταιρείες, π.χ. για μικρομεσαίες εταιρείες, οι απαιτήσει για αναφορά μπορούν να γίνουν ε, πιο ε, ελαφρές ή να είναι οι ίδιες σε διάφορους κανονισμούς. και θα ξεκινήσουμε αμέσως να ενσωματώνουμε κάποια από τα ευρήματά μας στις νομοθετικές προτάσεις που θα έρθουν σε ε, λίγους μήνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε είναι πολύ καλή η ερώτησή σας. Βεβαίως ε, ε, μην παρεξηγηθώ. Δεν πρόκειται εδώ πέρα για μια διάλυση του νομοθετικού μας που πρόκειται απλά για στοχευμένες παρεμβάσεις για να γίνει πιο αναλογικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως μπορούμε να ολοκληρώσουμε την πολύ επικοδομητική αυτή ανταλλαγή απόψεων και δάτω με τις ευκαιρίες να θέσω κάτι το οποίο είχε συγχωνευτεί στην συζήτηση του SSM που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Κάποια ζητήματα δηλαδή που ακριβώς ε, θίγονται για εξέταση από την Κομισιόν, η οποία ακριβώς ξεκίνησε τώρα τον πυλώνα 2 για μια θετική λύση για το δίλημα αυτό περί σαφήνειας της νομοθεσίας και βεβαίως τώρα υπάρχει και αυτό το θέμα του αποθεματικού, αλλά και το θέμα βεβαίως επικοινωνίας, της αποκάλυψης, της αγορές ε, και ακριβώς τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε εθνικές ε, αρχές των αγορών που ίσως εφαρμόζουν διαφορετικά τους ε, κανονισμούς, που έχουμε ένα κοινό πλαίσιο και θα ήταν νομίζω πάρα πολύ χρήσιμο και εδώ είναι το ερώτημά μου μήπως η ΕΣΜΑ και οι Κομισιόν μπορούν να συνεισφέρουν για μια ενιαία εφαρμογή αυτού του πυλώνα στην Ένωση και στην Τραπεζική Ένωση. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε τώρα. Αλλά προέκυψε από συζήτηση με την κυρία Νουή και συμφωνεί και αυτή ότι είναι ένα δύσκολο θέμα. Δεν ξέρω, θέλετε να απαντήσετε. Uh, uh, λοιπόν, απλά μια πολύ γρήγορη απάντηση. Για... Θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο της πρότασής μας, που θα αποτελέσει κομμάτι του νομοθετικής δέσμης μέτρων. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να κλείσουμε. Να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης και τους υπόλοιπους συναδέλφους που έχουν παραμείνει εδώ για να συζητήσουμε αυτό το του σημασία ζήτημα για την ε, αναθεώρηση του τραπεζικού τομέα. Θα έχουμε η ψηφοφορία για το ψήφισμα αύριο και θέλουμε να υπάρχει και συνοχή και με, την αρχή που με τις αρχές που παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης αφενός αντιμετωπίζοντας την ε, η υπερβολική βιωσιμότητα των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και τηρώντα και τι δεσμεύσει για μη υπερβολικές κεφαλαϊκές απαιτήσει και ίση συνθήκε ανταγωνισμού μεταξύ δικαιοδοσιών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε το διάλογο αυτό.